Good afternoon, everybody, dear colleagues. Καλησπέρα σας, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την ημερήσια διάταξη που πρέπει να εγκρίνουμε. Ελπίζω να μην έχετε καμία αντίρρηση. Ανακοινώσει του Πρόεδρου δεν έχουμε. Σημείο έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Έχει κάποιος κάποια αντίρρηση ή όχι. Ξεκινάμε λοιπόν με την ακρόαση για την κατάσταση στην ε, περιοχή των μεγάλων λιμνών. Θα γίνει από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Η κυρία Λέντα Μακάβαν είναι εδώ και θα συμπροεδρεύσει. Για Να αντιληφθούμε λοιπόν τις προκλήσεις αυτής της περιοχής. Καλωσορίζω τους δύο μιλητέ τον Δόκτωρα Ζεραρινιέ, ο οποίος είναι ερευνητή ε, στο κέντρο της Αφρικής ε, του Ατλαντικού Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Πατρίξ Κρυλέ, Διευθυντή Τμήματο ε, Κεντρική Αφρική στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και μέχρι πρόσφατα πρέσβη τη Ένωση στο Μπουρούντι. Όπω ξέρετε, υπάρχει μεγάλη ένταση στην περιοχή, πρώτα απ' όλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχει λήξει η εντολή του Πρόεδρου Καμπιλά και στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια κατάσταση εκτός συντάγματος, εφόσον δεν τροποποιήθηκε το σύνταγμα για να μπορέσει να έχει τρίτη θητεία. Ο κύριος Καμπυλά τώρα διακινδυνεύει το μέλλον της ε, χώρας του με ένα συνταγματικό πραξικόπημα καθώς σκοπεύει να καθυστερήσει τις εκλογές μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Η κατάσταση, η οποία είναι όλο ένα και πιο ασταθής, η βία, ο εκφοβισμός των πολιτικών αντιπάλων, των δημοσιογράφων και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανησυχούν ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο Υπενθυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μογκερίνη στην Ολομέλεια και εγκρίναμε και το σχετικό ψήφισμα. Το μέγεθος και μόνο της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό στην καρδιά της Αφρικανικής ε, Υπήρου και η αστάθεια της περιοχής δείχνει την ανάγκη που υπάρχει για μια αφρικανική και διεθνή αντίδραση. Στο γειτονικό Μπουρούντι, ο πρόεδρος Νουκουντσίζα επανεξελέγει για μια τρίτη θητεία τον Απρίλιο του 2015 και έκτοτε η χώρα βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση και από ό,τι φαίνεται πετεύχθη το αποτέλεσμα αυτό μέσω της άσκησης πίεσης ε, στο συνταγματικό δικαστήριο και μιας αναξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας. Είχαμε βία, 300.000 πρόσφυγες, κάποιοι μιλούν και για μια πιθανή γενοκτονία. Φαίνεται λοιπόν ότι επαναλαμβάνεται κάτι ανάλογο και στην Ρουάντα, όπου ο πρόεδρος Καγκαμέ σκοπεύει να κατεβεί για τρίτη θεία του 2017 μετά την αλλαγή και εκείνου του συντάγματος επιπλέον. Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες έχουμε τα γνωστά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνη με διασυνοριακές διαστάσεις και ελπίζω να αναφερθείτε σε αυτά στις ε, παρουσιάσεις σας ή στην συζήτηση. Τέλος. Φαίνεται πως η εξόριξη ορυκτών στο Ανατολικό Κονγκό σχετίζεται με το ότι κάποιε ένοπλε ομάδε βρίσκουν έτσι πόρου για να χρηματοδοτήσουν την σύγκρουση. Πριν από δύο εβδομάδε λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατέληξαν σε μια συμφωνία για τον κανονισμό για τα ορυκτά από έτσι ώστε ορυκτά και μέταλλα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξορίσονται με τρόπο υπεύθυνο. Θα δώσω λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Λίντα Μακάβαν, πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, για να πει δύο λόγια να έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο να υπάρξει παρακολούθηση της κατάστασης στις μεγάλες λίμνες της Αφρικής. Οτιδήποτε συμβεί εκεί θα έχει επιπτώσει στην σύνολη Αφρική. Είπατε κυρία Πρόεδρε ότι υπάρχουν διάφορες καταστάσεις δυσμενών εκλογικών συνθήκων. Υπάρχουν διάφοροι πρόεδροι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία και είχαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά μας για τη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό ζητήσαμε να εφαρμοστεί το άρθρο 26 και να κολλαστούν οι πράξεις ορισμένων στρατιωτικών που ασκούν καταστολή στο Κονγκό. Φυσικά έχουμε αναστείλει και την άμεση βοήθεια προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί εκεί μετά τις εκλογές. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη αστάθεια και στις δύο χώρες αυτές. Και με πρόσκληση του δόκτωρα Αντώνης Μουκουέβγε πήγα στο νοσοκομείο του στην, ε, στο Κονγκό που είναι ένα γενικό νοσοκομείο σε μια από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, αλλά ασχολείται ιδίω με γυναίκες οι οποίες είναι θύματα σεξουαλικής βίας, που πολλές φορές αυτό είναι και αποκοίημα των συγκρούσεων για ορυκτά σε εμπόλεμες ζώνες, στο Ανατολικό Κονγκό βέβαια, είναι και ο χώρος όπου έχουν μεταφερθεί όλα τα προβλήματα, ακόμα συνεχίζονται οι εντάσεις μετά από, την, ε, από τον εμφύλιο της Ρουάντα και ο δόκτωρ Μουκουέγγε είναι ένας πολύ θαραλέος άνδρας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε τη βία εκεί. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η ακρόαση και έχουμε επίση να αντιμετωπίσουμε και μια ανθρωπιστική κρίση γιατί όταν μιλάμε για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων που καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες. Έχουν φύγει 250.000 πρόσφυγες από το Μπουρούντι τους, τις τελευταίες εβδομάδες και πήγαν στη Ρουάντα. Με, πολλοί από αυτούς μετακινούνται τώρα προς την Τανζανία. Η κύληση αυτή ανθρώπων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αστάθεια και στην περιοχή των μεγάλων λιμνών <clears throat> λόγω της αντιπαράθεσης εθνοτικών ομάδων. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τα προβλήματα αυτά να πάρουν τη μορφή που είδαμε στην δεκαετία του 1990. Ήμουνα στο Μπουρούντι δύο εβδομάδες πριν από τις πρόσφατες ε, ταραχές και τότε μου λέγανε οι άνθρωποι ότι είμαστε μια ελληνική χώρα, ανησυχούσαν βέβαια για αυτό που θα συμβεί στις ε, εκλογές, αλλά δεν ξέραν τι θα συμβεί μετά από κάποιες εβδομάδες. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας και να ακούσουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει για να μπορέσει <clears throat> να αποτρέψει τη συγκρούσεις εκεί και να βελτιώσει την ανάπτυξη της περιοχής. Δίνω λοιπόν καταρχήν το λόγο στον κύριο Ζεραπρίνιε. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε ερωτήσει και απαντήσει. Μόλι ολοκλήρωσα μια έκθεση για έναν ε, πελάτη μα. Ε, ξέρετε ότι κάνω και consulting αυτές τις μέρες. Ε, όσον αφορά την στάση των όμορων χωρών όσον αφορά την, το μη σεβασμό των ε, συνταγματικών προθεσμιών ε, της προεδρικής θητείας από τον πρόεδρο Καμπίλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και είναι ιδιαίτερα αρνητικά από ό,τι φαίνεται τα πορίσματα. Κανείς δεν ασκεί πίεση όσον αφορά την τήρηση της προεδρικής αυτής θητείας και των σιωνικών ε, χρονοδιαγραμμάτων και νομίζω ότι η μόνη αν θέλετε επίκριση ήρθε από την πρόεδρο της Κεντροφρικανικής Δημοκρατίας που δεν έχει όμως επιρροή. Ήρθα σε επαφή με ηθήνοντε από τι όμορε χώρε και κανεί δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την τήρηση του συντάγματο όσον αφορά την προεδρική θητεία. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα απλώ να περιοριστώ στο ύφο τελικά τη ηγεσία που βλέπουμε σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε χώρε οι οποίε δεν υφίσταντο καν πριν από 50 χρόνια. Συνεπώς βρισκόμαστε σε μία τέταρτη αν θέλετε περίοδο αν θέλετε τώρα. Η πρώτη περίοδος ήταν απλώς η ε, περίοδος αμέσως μετά το τέλος της ε, απεικιοκρατίας. Ήταν ε, η περίοδος εκείνη κατά την οποία τα άτομα εκείνα τα οποία ήταν μέλη της, του εθνιστικού κινήματος κατά τη διάρκεια της απεικιοκρατίας είχαν στα χέρια τους την εξουσία. Ολοκληρώθηκε η περίοδος αυτή και πήγαμε σε μια περίοδο πραξικοπημάτων. Τη δεκαετία του 70 όλες οι χώρες αυτές πέρασαν από στρατιωτικά πραξικοπήματα. Ορισμένα από αυτά ήταν πάρα πολύ καταστροφικά όπως στην Ουγγάντα ή, που, ή του Μποκασά για παράδειγμα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Άλλα πάλι πραξικοπήματα ήταν πιο ήπια μπορούμε να πούμε. Πάντα Πάντως όλα είχαν αρνητικές επιπτώσεις, ορισμένα ήταν άκρο αριστερά, άλλα άκρο δεξιά και πολλές φορές είχαν να κάνουν και με τον ψυχρό πόλεμο εκείνης εποχής. Για παράδειγμα, το πραξικό μας στην Αιθιοπία είχε σαφώς ένα σοβιετικό προσανατολισμό και επηρεαστεί από τη Μόσχα. Κάθε πιθανή κατάσταση ουσιαστικά είχε προκύψει στα πλαίσια των πραξικομάτων αυτών. Το τέλος του ψυχρού πολέμου όμως έθεσε τέλος και σε αυτή την ευθυγράμμιση αν θέλετε. Όχι μόνο το να στρέφεται κανείς αριστερά ή δεξιά από πολιτικής πλευράς, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και αυτή η τάση των πραξικοπημάτων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, θα έλεγα ότι περάσαμε σχεδόν σε δημοκρατικές καταστάσεις και δημοκρατικούς θεσμούς. Ορισμένες χώρες ήταν αυθεντικά δημοκρατικές, όπως η Γκάνα, η Σενεγάλη, η Νότιος Αφρική, και αυτό μας προκανεί εντύπωση βέβαια, καθότι μόλις είχε τελειώσει το Απαρτχάιτ, αλλά ουσιαστικά αυτό οδήγησε στην ε, υφιστάμενη τέταρτη τρέχουσα περίοδο, όπου έχουμε μία σχεδόν δημοκρατική κατάσταση, μια κατάσταση σχεδόν δημοκρατικών βασιλείων θα τη λέγαμε. Οι ε, πρώην ε, επαναστάτες υπέρ της ελευθερίας έχουν γίνει τώρα βασιλείς. Και βλέπουμε ότι και σε άλλες χώρες, όπως και στην Γκαμπόν, ανάλογες τάσεις παρουσιάζονται. Στην πράξη λοιπόν, το καθεστώς ηγεσία αυτή τη στιγμή συνδέεται με την δυνατότητα να μπορεί κανείς να παραμένει περισσότερο στην εξουσία μέσω του συντάγματος, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική τήρηση του συντάγματος. Και ένα καταπληκτικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε με τον Ζώζεφ Καμπίλα, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος ήταν πρώην κομμουνιστής και ανήκε στην προηγούμενη περίοδο, όπου όπως σας είπα είχαμε αντιπαράθεση μεταξύ των φιλορώσων και αυτών που ήταν κατά των Ρώσων. Ουσιαστικά ήταν ένα έδος εκδίκησης για τον πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2001, σύντομα λοιπόν αφού είχε λάβει την εξουσία, και ο ευφυής λοιπόν αυτός, νεαρός εκείνη την εποχή, κατάλαβε τελικά να καταλάβει πάρα πολύ καλά τι θα έπρεπε να κάνει ότι θα έπρεπε δηλαδή να κάνει ότι είναι δημοκράτης χωρίς την πραγματικότητα να είναι δημοκράτης. Και αυτή τη στιγμή βασικά έχουμε μία τρίπτυχη θα έλεγα αντιπαράθεση εξουσίας. Η μία πτυχή, η μία πλευρά και παραθατικά σας λέω εδώ πέρα ότι θα ήθελα να χαιρετήσω την μνήμη του Μάλι Μουνιερερέ που ε, μετά την ε, εισβολή του 1978 πήγε στην Αντίσα Μπέμπα και είπε ότι χρειάζεται βοήθεια κατά της ξένης εισβολής. Και του είχαν πει τότε ότι ο, ο Δόκτωρ Μπεντζαμίν ήταν πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμεί τέτοια αρνητικά πράγματα, του είχαν πει. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που ήταν πάρα πολύ ειλικρινής, εκνευρίστηκε πάρα πολύ και είπε όχι, εσείς δεν είστε πραγματικά μια οργάνωση Αφρικανικής Ένωσης, ίσως αστικά μια συνδικαλιστική οργάνωση επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Και συμφωνώ ουσιαστικά με την προσέγγιση αυτή. Λοιπόν, μία πτυχή, αν θέλετε, της αντιπαράθεσης εξουσίας που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς η συνδικαλιστική οργάνωση επικεφαλής κρατών κυβερνήσεων που, είχε, που έχει προκύψει. Και ουσιαστικά είναι πολύ πιο νοσηρή από ό,τι ήταν το 1978. Και αυτό γιατί η διεθνής κοινότητα έχει ενδυναμώσει τους αρχηγούς αυτούς κρατών και κυβερνήσεων με έναν τρόπο που δεν μπορούσε καν να τους υποστηρίξει το 1978, ακριβώς επειδή τότε είχαμε τον ψυχρό πόλεμο. Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με τους ε, ανθρώπους που κατεβαίνουν στο δρόμο. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις που έδωσε η Δύση για τη δημοκρατία, για το ότι θα πρέπει ουσιαστικά να έχουν όλοι πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες ε, όσον αφορά τα δημοκρατικά καθεστώτα. Ακριβώς ε, αυτό το έλαβαν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί πολίτες. Όταν θα φερθούμε σε λίγο στον Μπουρούντι θα καταλαβαίνουμε εκεί πέρα ότι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στους δρόμους και η αστική τάξη δεν είναι τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός, ο πρόεδρος του Μπουρούντι, εξελέγει δημοκρατικά, ότι θεωρείται ότι η τελευταία αυτή εκλογή του δεν ήταν ε, συνταγματική, έλαβε παρόλα αυτά ένα 65%. Εντάξει, γίνανε κάποιες μικρές νοθείες όσον αφορά, αλλά τίποτα το τόσο όσον αφορά την εκλογή του, τίποτα τόσο σοβαρό. Όταν λοιπόν τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο, δρόνο, στο δρόμο, Αναφέρω, αναφέρομαι στους ανθρώπους εκείνους που κατοικούν στις πόλεις, που είναι η μειοψηφία τελικά αυτή από ό,τι συμβαίνει στη Δύση, από ό,τι συμβαίνει στην Ασία, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά κατοικούν πλέον στις πόλεις και είναι ελάχιστοι στην Ήπεθρο. Στην Αφρική συμβαίνει το αντίστροφο. Επομένω θα έλεγα ότι η δημοκρατία αποτελεί αυτή τη στιγμή όνειρο για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους και οι οποίοι κατοικούν στις πόλεις. Δεν λέω ότι δεν ονειρεύονται τη δημοκρατία και άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα για αυτούς όσο είναι για τους ανθρώπους που κατοικούν στις πόλεις. Και η τρίτη πτυχή είναι εσείς ουσιαστικά, η διεθνής κοινότητα. Η δική σας άποψη, η δική σας στάση γίνεται αντιληπτή από τις χώρες αυτές. Ορισμένες φορές επικρίνεται, άλλες φορές δημιουργεί και εμφυσά ελπίδα, αλλά σαφώς η δική σας συστάση έχει θετική ή αρνητική επίπτωση. Έχει αντίκτυπο ο λόγος σας. Ο αντίκτυπος βέβαια τώρα αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά αντίκτυπος πάντα υπάρχει. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές πτυχές τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις όσον αφορά τον αγώνα αυτό που γίνεται για την ανάκτηση της εξουσίας. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στον δρόμο, οι απλοί πολίτες που ζουν στις πόλεις, η άποψη της διεθνούς κοινότητος και από την άλλη αυτό το οποίο εγώ αποκαλώ τα συνδικάτα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, που ουσιαστικά δεν αφουγκράζονται τους πολίτες των χωρών τους, διαφορετικά θα είχαν μια πιο δημοκρατική στάση. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και το Κονγκό επίση δεν είναι μόνο η περιοχή των μεγάλων λιμνών, επηρεάζει την Κεντρική Αφρική και τη Δυτική Αφρική. Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θα έλεγα ότι είναι μια τεράστια χώρα, μια τεράστια επικράτεια στην καρδιά πραγματικά τη Αφρικανική Υπήρου και δεν νομίζω ότι μπορούμε απλώ να κατατάξουμε τη χώρα αυτή σε μία μόνο κατηγορία όπω οι μεγάλε λίμνε. Επηρεάζει και πολλέ άλλε περιοχέ τη Αφρική. Με την άδειά σας λοιπόν κυρία Πρόεδρε και θα ακούσουμε και τον άλλο συνάδελφο, θα ήθελα ή δυνατόν να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά τη θέση συγκεκριμένων χωρών για την κατάσταση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, για την Μπραζαβίλ, η Ρουάντα, η Καμπάλα ή την Μπουζουμπούρα δεν έχουν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα αυτή. Ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο. Thank you. Thank you, doctor. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ε, αναμένουμε βεβαίω και τις ερωτήσεις. Το κύριο Σπίρλε. Θα ακούσουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική κρίση και στην κρίση ασφαλείας, η περίπτωση του Μπουρούντι. Έχει τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μου ζητήσατε να πάρω το λόγο και να σας μιλήσω για την περιοχή των μεγάλων λιμνών της Αφρικής. Το τέλος της α, επανάστασης των M23, η υπογραφή της α, συμφωνίας στην Αντίσα πραγματικά μας έδωσε την ελπίδα ότι όντως θα υπήρχε πλέον η δυνατότητα σταθεροποίησης στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Δυστυχώς όμως οι εθνικές κρίσεις τελικά δεν το επέτρεψαν αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ στην κατάσταση που επικρατεί τόσο στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά πιο ιδιαίτερα στην κατάσταση που επικρατεί στο Μπουρούντι. Θα έλεγα ότι είναι δύο κρίσει που απασχολούν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι οποίε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε πραγματικά να συμβάλλει για την επίλυσή του. Όσον αφορά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, όλοι γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία τη 19η Δεκεμβρίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Τότε ολοκληρώνεται η προεδρική θρητεία του Καμπίλα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τρέχει ο χρόνο, πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο, ακούμε αντικρώμενε πληροφορίε μέχρι να φτάσει αυτή η ημερομηνία και από ό,τι φαίνεται υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επαναδιαπραγμάτευση με τη συμμετοχή της ε, ΣΕΜΚΟ. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μια συμφωνία του Οκτωβρίου όσον αφορά την ε, συμβολή τη Αφρικανικής Ένωση. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ήδη μια επίκριση όσον αφορά τη δυνατότητα διαμεσολάβησης και από ό,τι φαίνεται θέλουν αυτή τη στιγμή να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθούν να δουν αν τελικά θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία βάσει της πρότασης της ΣΕΜΚΟ και βάσει της συμφωνίας της 18 Οκτωβρίου. Καθότι όμως προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βρουν μια διαβριμένη λύση, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι σταθερή και ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι. Η είπατε εκπρόσωπος το είπε πριν από λίγο καιρό ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτον, είπε ότι ε, η συμφωνία της 18 Οκτωβρίου θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση, αλλά δεν αρκεί από μόνη τη και θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να είναι πιο ανοιχτή προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την Προεδρία του κυρίου Καμπίλα μόνο βάσει συμφωνίας αυτή, πέρα από 19 Δεκεμβρίου θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτό. Η χώρα αυτή γνωρίζει στα ανατολικά της κυρίως μια παρατεταμένη κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν να περάσει αυτή τη στιγμή από μια επέκταση προεδρικής θητείας η οποία ενδεχομένω να ενέχει και τον κίνδυνο περισσότερων συγκρούσεων. Θα πρέπει σαφώς εφόσον παραταθεί η θητεία του κύριου Καμπίλα να υπάρχουν και επιπλέον μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να κατευνάσουν τον κόσμο όσον αφορά για παράδειγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τους πολιτικούς κρατούμενους ή όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην αντιπολίτευση και τα αντιπολιτευόμενα πολιτικά κόμματα. Η παράταση αυτή της προεδρικής θητείας του κ. Καμπίλα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομη και ουσιαστικά να επιτρέψει το συνδυασμό των προεδρικών, των ε, βουλευτικών και των τοπικών εκλογών. Τέταρτον, η δέσμευση του ίδιου του Ζωζεφ Καμπίλα ότι δεν πρόκειται να υποβάλει εκ νέου αίτηση, υποψηφιότητα για το προεδρικό αξίωμα. Θα πρέπει αυτό να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας και θα πρέπει αυτό ουσιαστικά να λειτουργήσει ως μέτρο το οποίο θα ευνοήσει την συμφιλίωση. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπατε εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε κάποιες ανησυχίε όσον αφορά το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφερόμενοι πιο συγκεκριμένα στις ε, πολύ ε, άσχημες εικόνες που είδαμε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σεπτεμβρίου, που 50 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και όπου ε, είδαμε ότι υπήρχαν έντονα φαινόμενα καταστολής, τα οποία επέκρινε το Κέντρο Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσει και περιοριστικά μέτρα όσον αφορά του ηθήνοντε για τα μέτρα αυτά καταστολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω πέρα από την ίδια την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνής κοινότητας και οι ίδιοι εταίροι της περιοχής αυτής να συμβάλλουν περισσότερο, ιδίω όσον αφορά τη συμβολή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και εδώ ουσιαστικά τα όσα λέω συνδέονται και με αυτά που είπε πριν από λίγο ο κύριος Πχουνιέ. Η Αφρικανική Ένωση και οι όμορε χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειε, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει μια γενικότερη αποσταθεροποίηση σε όλη την περιφέρεια. Ορισμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τη περιοχή αυτή ήδη έχουν αναλάβει δράση. Τα Ηνωμένα Έθνη επίση μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο, λαμβάνοντα ιδίω υπόψη την ξεκάθαρη θέση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 77 όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια και το άλλο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί για τι προεδρικέ εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχυθεί ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ηθήνοντες στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βάσει του άρθρου 8 και σύμφωνα με τη Συμφωνία του Κοτονού προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη χώρα αυτή προκειμένου να αρχίσει να ακολουθεί συγκεκριμένες δημοκρατικές αρχές και ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο προτεραιοτήτων πολιτικών. Είναι σημαντικό να γίνει μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, των αστυνομικών αρχών και μεταρρύθμιση του γενικότερου τομέα της ασφάλειας. Και αυτά αποτελούν ε, τμήμα του ενδεικτικού προγράμματο της ανδεξιακή Βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Πρέπει επίσης να καταβληθούν οι απαραίτητε προσπάθειες προκειμένου να δούμε πώς θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε την, ε, δημοκρατία, την ε, διαδικασία εκδημοκρατισμού και πώς τελικά θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια εκλογική επιτροπή η οποία θα είναι σταθερή και η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Τόσα συμβούν τι επόμενε εβδομάδε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εκ του σύνεγγυ να παρακολουθεί την κατάσταση και θα πρέπει να υποστηρίξει τις προτάσεις της ΣΕΜΚΟ, καθώς επίσης και κάθε πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της εμπιστοσύνης, μάλλον σε μείωση της έλλειψης εμπιστοσύνης που υπάρχει αυτή τη στιγμή και προτού φτάσουμε στην ημερομηνία της, του τέλους Δεκεμβρίου. Και θα πρέπει ο Πρωθυπουργό τώρα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η α, κυβέρνηση που θα σχηματίσει να έχει την α, γενικότερη συνένεση των εμπλεκόμενων μερών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να προσέξει πάρα πολύ την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και αυτό πρέπει να γίνει και με τη συμβολή των υπόλοιπων διεθνών εταίρων. Όσοι είναι υπεύθυνοι για την βίαιη καταστολή θα πρέπει να αποτελέσουν, ε, αν θέλετε, τους πρώτους στόχους των ε, στοχευμένων αυτών περιοριστικών μέτρων που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όσον αφορά την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Θα ήθελα τώρα με την άδειά σας να αναφερθώ και στο Μπουρούντι. Όπως ακούσατε, ολοκλήρωσα πριν από λίγο την θητεία μου ως πρεσβευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή και θα έλεγα ότι αξίζει εδώ πέρα να κάνουμε μία σύγκριση με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ πέρα έχουμε μία ιδιαίτερη, αν θέλετε, πορεία και νομίζω ότι θα πρέπει ξεχωριστά να εξετάσουμε τις δύο αυτές χώρες. Είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η όλη βάση και από πηγάζει η κρίση, η πολιτική διάσταση τη κρίση αυτή, η διάσταση που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την κοινωνία, την οικονομία, τι εθνοτικέ ομάδε, καθώ επίση και τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιληθεί η κρίση. Όσον αφορά τα βασικά αίτια τη κρίση αυτή, πού βασίζεται αυτή η κρίση. Σαφώ υπάρχουν πολύ πιο ειδήμονε από μένα για να απαντήσουν στο ζήτημα αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα σε ορισμένα στοιχεία να επιμείνω χωρίς να επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πρώτο σημείο. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παρακαταθήκη που έχει αφήσει η ιστορία. Αναφέρομαι στην περίοδο από το 1972 και μετά, μέχρι το 2014, καθώς επίσης και με την δολοφονία του Πρόεδρου Αντάι. Πώς μπορούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε την ε, άποψη που έχει αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη όσον αφορά τον πρόεδρο Νουκουρουνζίζα και πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσεγγίσουμε όλες αυτές τις ομάδες ανταρτών που αντιβαίνουν στην ε, κυβέρνηση και τέλος να δούμε πώς αντιμετώπισε η φυστάμενη κυβέρνηση την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε πριν από λίγο καιρό και ποια είναι η υποστήριξη που δίνει η κοινή γνώμη προς το πραξικόπημα αυτό. Το ΣΕΝΕΦΔΕΝΤΕ, το οποίο είναι το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται θέλει να παραμείνει στην εξουσία, αλλά θέλει ουσιαστικά να πάρει και μία εκδίκηση σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα στον Μπορούντι. Και αυτό το είδαμε και πρόσφατα. Μέσω της διαδικασίας αυτής περαιτέρω εγκατάσταση στην εξουσία του κυρίου Κουρουνζίζα με μια συνεχή αποδυνάμωση των αντιπολιτευτικών πολιτικών κομμάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της προκλογικής περίοδου. Δεύτερο τώρα σημείο, η πολιτική διάσταση της κρίσης. Όπως το ξέρετε έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες διαλόγου αυτή τη στιγμή στον Μπορούντι. Μια διαδικασία σε εθνικό επίπεδο και μια διαδικασία σε περιφερειακό επίπεδο υπό την αιγίδα της ε, ανατολικοαφρικανικής κοινότητας. Όσον αφορά τον εθνικό διάλογο που προωθεί η εξουσία, προφανώς αυτός δεν περιλαμβάνει τους πάντες. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν και η βασική ανησυχία ως προς το διάλογο αυτό είναι ότι ε, τα πορίσματα του διαλόγου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τελικά για την μεταρρύθμιση του συντάγματος και για την ε, διαιώνιση τελικά του υφιστάμενου Προέδρου στην εξουσία δημιουργώντας τη δυνατότητα να παραμείνει ο άνθρωπος αυτός στην εξουσία για πάνω από δύο θητείες. Και μάλιστα η δικασία αυτή ήδη έχει ξεκινήσει. Και προβλέπεται ακόμα και η δυνατότητα χρησιμοποίησης δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συντάγματος. Σε περιφερειακό επίπεδο επίσης δεν προχωράει ο διάλογος. Ο κύριος Μοκαπέ που είναι ο διαμεσολαβητής για τον περιφερειακό αυτό διάλογο είπε ότι μέχρι το 2017 ολοκληρώνεται η θητεία του. Από τη μία όμως πλευρά έχουμε τις ομάδες εκείνες, τις αντιπολιτευτικές, οι οποίες έχουν χάσει πλέον την εμπιστοσύνη τους απέναντι στο διάλογο αυτό και άρα σιγά σιγά ενδεχομένω να αναλάβουν πάλι η δράση και από την άλλη έχουμε το κυβερνών κόμμα το οποίο δεν μαλακώνει τη στάση του, ιδίως όσον αφορά τον κατάλογο αυτό αποκλήσεων δηλαδή τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτικών κομμάτων και όλων των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στον εθνικό περιφερειακό αυτό διάλογο, καθότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα περισσότερα από τα κόμματα αυτά ως συνδεδεμένα με την απόπειρα πραξικοπήματος. Επόμενη διάσταση τώρα του ζητήματος ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Η διάσταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ουσιαστικά θα έλεγα ότι αυτή που προκαλεί και τις περισσότερες ανησυχίες. Πληθώρα εκθέσεων αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί από το Human Rights Watch, από άλλους οργανισμούς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΕ όσον αφορά την ανησυχητική κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Μπουρούντι. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συνεχής άρνηση αναγνώρισης της ανησυχητικής κατάστασης από την κυβέρνηση του Μπουρούντι. Τα αριθμητικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα σοκαριστικά. Έχουμε εξαφανίσεις, βασανισμούς, εξοδικαστικές εκτελέσεις, καθώς επίσης και ομαδικές ενταφιάσεις μετά τα γεγονότα του 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί βέβαια τις παραβιάσεις αυτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οποιοδήποτε και αν είναι ο υπεύθυνο. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Επίσης, ας δούμε λίγο την κοινωνικο-οικονομική διάσταση της κρίσης. Ξέρετε ότι το Μπουρούντι κατά 50%, ο προπολογισμό του κατά 50% εξαρτάται από την εξωτερική βοήθεια μέρος της οποίας ε, ανεστάλλει και επανα, πρόσφατα και κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός πληθυσμού που είναι πάρα πολύ φτωχός. Έχουμε ήδη μια έντονη ανθρωπιστική κρίση, ας δούμε τους ε, δείκτες υποσυτισμού για παράδειγμα για τη χώρα και μόνο η τεράστια τελικά ανθεκτικότητα του πληθυσμού μειώνει κάπως ε, την εμβέλεια των αρνητικών αυτών επιπτώσεων. Επίσης βλέπουμε ότι εξαφανίζονται όλο και περισσότερο κάποιες βασικές υπηρεσίες ε, δημόσιες από τον Μπουρούντι, ότι οι υπηρεσίες αυτές είχαν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από τη διεθνή κοινότητα. Και επίσης βλέπουμε ότι μειώνεται η δυνατότητα του κράτους αυτού να αντιμετωπίσει την κατάσταση, καθότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανώτεροι εξωματούχοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα αυτή και δεν μπορούν πλέον να συμβάλλουν σε προσπάθειε ανοικοδόμηση. Α μην ξεχνάμε ότι έχουμε περίπου 300.000 ανθρώπου που είναι πρόσφυγε σε γειτονικέ χώρε. Η κρίση όμω στον Μπουρούντι έχει και μια εθνοτική διάσταση. Και αυτό διότι βασίζεται σε μια ιστορική πραγματικότητα για τη χώρα αυτή και από την άλλη γιατί υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη πόλωση όσον αφορά συγκεκριμένε ελίτ. Ορισμένε δηλώσει και διακηρύξει του κυβερνώντο κόμματο ουσιαστικά έχουν τροφοδοτήσει την πόλωση αυτή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει εδώ πέρα να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, η πολιτική αυτή αντιπαλότητα για την κατάκτηση εξουσίας φέρνει σε αντιπαράθεση μεταξύ τους και τις ίδιες τις ε, παρατάξεις Χούτου, FNL και Φροντεμπού για παράδειγμα. Και νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης και το γεγονός ότι ε, ορισμένοι παράγοντες Τούτσι ουσιαστικά συνδέονται αυτή τη στιγμή με την ε, κυβέρνηση που ε, με το κυβερνον κόμμα. και την κατάσταση όμως, μιλάω για την τρέχουσα κατάσταση, εξακολουθεί να παρουσιάζει κινδύνους, ιδίως λόγω των ρογμών που έχει δημιουργήσει σε εσωτερικό επίπεδο στις δυνάμεις τάξης. Και αυτά για να σας ε, παρουσιάσω την κατάσταση στην τελευταία αυτή πτυχή. Ποια είναι τώρα η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα εμείς θα πρέπει να αντιταχθούμε προφανώς και να ζητήσουμε να υπάρχει μια περιφερειακή και ακόμα παναφρικανική λύση. Τα γεγονότα δείχνουν ποια είναι και τα όρια μιας τέτοιας προσέγγισης παρά τις ε, φιλότιμες προσπάθειες του πρώην Πρόεδρου Μουκαπά. Συγχρόνως θα πρέπει να υπάρξει Συντονισμό των προσπαθειών μας μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Τη στιγμή όμως που η κυβέρνηση του Μπουρούντι κάνει συστηματικές προσπάθειες να αποδυναμώσει το ρόλο του ΟΗΕ. Παραδείγματο χάρη, άρνηση να συζητήσει με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών, <clears throat> άρνηση συζήτηση των προτάσεων που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πιο πρόσφατα η άρνηση να υπάρξει παρουσία του, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Και αυτό ακολουθεί την ε, προκατακτική έρευνα κατά του Μπουρούντι που έχει ξεκινήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσει τις προσπάθειές σας για να υπάρξει μια διαβούλευση βάσει του άρθρου 96 για τα κατάλληλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε περαιτέρω, θέλω να υποχρεωθήσω όμω τα εξή. Εδώ. Πρώτα απ' όλα, είμαι πεπισμένο ότι το άρθρο 96 και η εφαρμογή του είναι απόλυτα δικαιολογημένη τη στιγμή που δεν έχουν τηρηθεί τα υπεσχημένα σε επίπεδο εταιρική σχέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατικοποίηση στον Μπουρούντι. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι δεσμεύσει οι οποίε θα πρέπει να εκπληρωθούν από την πλευρά του Μπουρούντι απαιτούν μία πολιτική θέληση και μόνο και ανοιχτό πνεύμα. Οι προσδοκίες που υπάρχουν για διάλογο, οι προσδοκίες για την ανεξαρτησία των μέσων ε, ενημέρωσης και των δικαστικών αρχών είναι βασικά στοιχεία αυτών των προσπαθειών. Και εξάλλου η, ο στόχος των διαβουλεύσεων δεν είναι να πάρουμε μέτρα κατά του πληθυσμού του Μπουρούντι που πρέπει να συνεχίσουμε να τον υποστηρίζουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά <clears throat> την προσέγγιση του άρθρου 96. Συγχρόνως έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων υπευθύνων για τις ομότητες που έχουν λάβει η χώρα και εναντίον αυτών οι οποίοι αντιτίθενται σε μια πολιτική λύση. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία της προσέγγισης της ευρωπαϊκή Ένωσης με την προσπάθεια να υπάρξει μια διευρυμένη πίεση της διεθνούς κοινότητας για διάλογο με την διαμεσολάβηση της κοινότητας Ανατολικής Αφρικής και με το άρθρο 16 και με τα περιοριστικά μέτρα εναντίον ορισμένων ηθινόντων. Για να κλείσω για το Μπουρούντι. Ε, πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι παραμένει μια στάση εμπλοκής υπάρχουν λύσεις. Με μια επιζήτηση μιας περιεκτικής πολιτικής λύσης αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε και εδώ θα ήθελα να κλείσω να υπάρξουν ελάχιστα μέτρα καταπράγηση τη κατάσταση από την κυβέρνηση και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μας, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Βάουτμανς που είχε ζητήσει την ακρόαση. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο κυρίους ε, για τις ε, παρουσιάσεις τους. Φαίνεται ότι είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, βλέποντας εδώ πέρα και την προσέλευση των συναδέλφων, αλλά νομίζω πως θα πρέπει λίγο να τα δει αυτά η Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε μια σχετική συνεδρίαση, μιλήσαμε με την κυρία Μογκερίνη για το Κονγκό, εγκρίναμε και ένα ψήφισμα και την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ, εδώ, στις Βρυξέλλες, ε, περνάει ο χρόνος, ε. εδώ ήταν στην Ολομέλεια των Βρυξελών που ψηφίσαμε το ψήφισμα για το Κονγκό και το ότι ο Καμπιλά παρατείνει την θητεία του. Εγώ γνωρίζω αρκετά καλά την κατάσταση που την Ρουάντα μετά την γενοκτονία. Είμαι νομίζω μία από τους λίγους ανθρώπους που είδα όλα αυτά τα κουτιά γεμάτα χέρια, πόδια, κρανία και πραγματικά αν θέλει κανείς να καταλάβει το τι συμβαίνει τώρα στο Μπουρούντι και το πώς ξεκίνησε η υπόθεση αυτή με την γενοκτονία θα πρέπει να ξέρει αυτά τα πράγματα και ανησυχώ πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι στο Κονγκό η κατάσταση είναι πάρα πολύ έφλεκτη και υπάρχει ο κίνδυνος πραγματικά να αναφλεγεί. Αν δούμε τις χώρες χωριστά, αν δούμε το τι συμβαίνει στο Κονγκό, πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος τώρα όντως να υπάρξει μια ανάφλεξη. Είχε βγει ο κόσμος στους δρόμους ε, και έλεγε καμπυλά, Λεφινή κτλ. Αν δούμε και το Μπουρούντι, έχω και εκεί πέρα φίλους και στους οποίους είχα μείνει και εκεί πέρα πραγματικά βλέπει κανείς πόσο άσχημα είναι οργανωμένα τα πράγματα και θα ήθελα να μου πούν και οι δύο κύριοι τελικά τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Μας είπατε εκεί πέρα, κοιτάει κανείς την περιοχή, την Αφρικανική Ένωση. Εμείς έχουμε εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνουμε πολλά λεφτά ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, εντάξει, ψηφίσματα δεν σημαίνουν τίποτα εκεί πέρα για τους ανθρώπους. Οπότε η πραγματική μου ερώτηση είναι αυτή. Όταν ισχύει κάποιος όπως εγώ και το κόμμα μου για την περιοχή, τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε πρέπει να καταλάβει ο Καμπιλά ότι θα υπάρξουν κυρώσεις, ε, θα υπάρξει απαγόρευση βίζας, θα παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα, αλλά πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Δεν μπορούμε ως Ευρώπη, ως παγκόσμια δύναμη να καθόμαστε και να κοιτάμε. Βιάζονται άνθρωποι καθημερινά στο Ανατολικό Κονγκό. Είχα πάει στο Κίβου και πραγματικά μιλήσαμε τα θύματα εκεί πέρα τα κοριτσάκια που βιάζονται και υπάρχει η κατάσταση αυτή χρόνια. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε να σταματήσει. Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα λέγατε, τι θα ζητούσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βόιτμαντς. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν αρκεί το να εγκρίνουμε ψηφίσματα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις των ε, εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Ο κύριος ε, Σαφχάζων είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρινιέ και τον κύριο Σπιλέ, ιδιαίτερα τον κύριο Πρινιέ, δείξατε πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα, γιατί πολλές φορές μέσω του, των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολλοί με καθαρή τη συνείδησή τους προσπαθούν να απλοποιήσουν μέχρι επίπεδου γελιογραφίας μια πολύπλοκη κατάσταση. Εγώ είχα βρεθεί ως εκπρόσωπος της χώρας μου στην ε, ε Γκόμα ε, όταν ε, εργαζόμουν με την μεταβατική κυβέρνηση. Τώρα, θέλω να πω κάτι και αυτό δείχνει λιγάκι περισσότερο το γενικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Είχαμε μία αυτήν την, αυτό το εγχείρημα του Λοράν Καμπιλά στο Κονγκό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά το διοργάνωσε απόλυτα από την αρχή στο τέλος μια εξωτερική ισχύς, μια εξωτερική δύναμη η οποία θέλησε να χρησιμοποιήσει τον Λοράν Καμπίλα για να αναχαιτήσει τους αντάρτες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Κάτι άλλο πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι μέσα σε, στο εγχείρημα αυτό εναντίον του Λοράντε Ζήρε Καμπιλά ο οποίος εμποδίστηκε από μια παρέμβαση της Γαλλίας από την Αγγόλα όταν ο Λοράν Καμπιλά θέλησε να στραφεί εναντίον αυτών που είχαν δημιουργήσει αυτήν την ε, αποσταθεροποίηση υποστηρίζοντας τους ε, αντάρτες εδώ στις Βρυξέλλες και ήμουν εδώ παρόν επάρθη, ελήφθη η απόφαση να δολοφονηθεί ο Λοράν Καμπιλά με την έγκριση του μεγάλου αδερφού, δηλαδή των ΗΠΑ. Όλα αυτά γεγονότα είναι πραγματικά στοιχεία. Είναι μια ιστορία που είναι μυστική, αλλά είναι μια πραγματική ιστορία που εγώ την έχω γνωρίσει από μέσα. Στη σημερινή κατάσταση λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή όχι μόνο αποσταθεροποιείται, μιλάμε για εκατομμύρια νεκρούς, 7 ή 8 εκατομμύρια. Και συγκρίνεται το αυτό με όλη τη φασαρία που κάνουμε για τη Συρία. Έχουμε 250.000 νεκρούς στη Συρία, 8-9 εκατομμύρια εκεί, λόγω εξωτερικής αποσταθεροποίησης στο Κονγκό. Όταν τα λέμε λοιπόν αυτά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Τι θέλω να πω. <clears throat> Ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο ο οποίος είναι περιεκτικός. Προφανώς να ακολουθήσουμε την πρόταση των επισκόπων για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο στο χρόνο. Και αυτό το σύνταγμα είναι τελείως νοπό θα πρέπει να δούμε πώς θα οικοδομήσουμε μια πραγματική μετάβαση και πώς θα επανέλθουμε και πάλι σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό εγώ ζητώ από το Κοινοβούλιο μας να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία μετάβασης με όλη τη δυνατή επιφυλακτικότητα. Τώρα, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση για να μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο σε αυτό το περιεκτικό διάλογο χρειάζεται ένα πραγματικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Όχι 50 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια. Ένα δισεκατομμύριο τουλάχιστον για αυτή την περιοχή που χρειάζεται ανάπτυξη και αν το κάνετε αυτό, εάν υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό σχέδιο Marshall για την περιοχή των μεγάλων λιμνών, μόνο έτσι μπορείτε να ξαναφέρετε Διαδικασίε, περιεκτικές και διαδικασίε ειρήνευσης. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, εάν θέλει να είναι πραγματικό παίκτη στην περιοχή. Και είναι εφικτό. Είναι δυνατό να κάνουμε τέτοιο πρόγραμμα με την υποστήριξη τη Παγκόσμια Τράπεζα ή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανάπτυξη. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τα πράγματα στην Αφρική, αυτό πρέπει να κάνουμε γιατί αλλιώ οι προσπάθειές μα μπορεί να αποσταθεροποιήσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Εγώ ήμουνα τότε που ήμουν στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, ερχόντουσαν οι μαφιόζοι ή τα ισλαμικά κυκλώματα, ερχόντουσαν με χρήματα και ξαναφεύγανε με χρυσάφι και διαμάδια. Αυτή η ζώνη είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για εμπόλεμες συνθήκες στον κόσμο. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι, αυτό είναι στο χέρι μας. Και αυτό μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο αντί να δίνει απλώς διδάγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βορείως της λαϊκής δημοκρατίας στο Κονγκό υπάρχει η, λαϊκή, η δημοκρατία του Κονγκό που δεν είναι λαϊκή. Εκεί πέρα κύβερνα ο ίδιο άνθρωπο 26 ε, χρόνια, ετοιμάζεται για την επόμενη επταετή θητεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως, δεν υπάρχουν εκατομμύρια νεκροί στο μη δημοκρατικό κόμπο. Και ίσως πρέπει να δεχτούμε το ότι ο εκδημοκρατισμό φταίει για την αποσταθεροποίηση αυτή. Ίσως πρέπει, δεν ξέρω, να πούμε στον κύριο Καμπυλά να γίνει ε, βασιλιάς ε, του Κονγκό ή ο βασιλιάς των Βέλγων να ξαναγίνει μονάρχης ε, του Κονγκό, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Αφρική. Σας ευχαριστώ. Η συμπρόεδρος, η κυρία Λέντα Μακάβαν τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρινιέ. Μου άρεσε αυτό το οποίο είπατε ε, μιλήσατε για κύματα της ιστορίας, ε, πράγματα συμβαίνουν, ξαναλάζουν και είπατε ότι ε, τελειώνει η εποχή του εκδημοκρατισμού. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι θα έχει η επόμενη εποχή και αν θα το δεχτεί ο κόσμος, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, το είπαν και αρκετοί συνάδελφοι. Ναι, εντάξει, εμείς ψηφίζουμε διάφορα πράγματα, λέμε εκεί πέρα διάφορα άρθρα, το άρθρο 96, κάνουμε δηλώσεις, αλλά... Αλλά δεν μας δίνουν και πολύ σημασία. Τι πρέπει να ζητάνε τώρα, να ζητήσουν οι διεθνείς οργανισμοί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ρουάντα, το και αν δεν αντιδράσουν, γιατί είμαι και Πρόεδρο τη Επιτροπής Απασχόληση, Μήπω να κόψουμε την βοήθεια αντί να γίνει ένα τεράστιο σχέδιο Μάρσαλ για το Κονγκό. Εκεί πάει η συζήτηση. Γιατί αν συνεχίσουμε να λέμε θα κάνουμε κάτι και μετά δεν κάνουμε, ε, μετά δίνουμε και την εικόνα κάποιου αδύναμου. Και οι υπόλοιπε δυνάμει ε, τώρα εκεί, ο κ. Σαφχάζο ανέφερε την Αλκάιντα, τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Οι υπόλοιπε δυνάμει ποιε είναι και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και λιγότερη συμμαχία. Τέλο, όλε αυτέ οι χώρε δεν είναι ίδιε όπω είπατε. Διαφορετικέ χώρε, διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν και αυτό για το οποίο πάντα με ρωτάνε είναι η Ρουάντα είναι ένα καλό παράδειγμα χώρα όπου ε, ο πρόεδρο λέει ότι θα είναι ξανά υποψήφιο για εκλογές, αλλά όπως είπατε, δεν είναι ότι θέλει και να το ξεφορτωθούν κιόλα από την ε, Ρουάντα, γιατί λαμβάνει πολύ ψηλά επίπεδα διεθνούς βοήθειας, γιατί τα πράγματα βελτιώνονται, η κατάσταση βελτιώνεται. Μήπως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν πρέπει να λέει να φεύγουν πρόεδροι σαν τον Καγκάμι άμα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στη χώρα τους. Με ρωτάνε για τέτοια πράγματα κάθε μέρα και θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη. Ξέρω πως ο κ. Πυρλέ βεβαίω θα εκφράσει την άποψη της Ένωσης, αλλά έχει οπωσδήποτε και μεγάλη εμπειρία στα ζήματα της Αφρικής, οπότε θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ευχαριστώ. Και εμένα η δικιά μου ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση πάει, γιατί μιλάμε για ψηφίσματα, για δηλώσεις, ε, και όπως είπε και ο Σαφχάουζερ, αποθελώ συγκεκριμένα μέτρα. Τι είπε και ο κύριος Βάτμας. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα ως διεθνή κοινότητα. Τι είναι η καλύτερη απάντηση. Πριν σας δώσω τον λόγο, θα ακούσουμε την Κομισιόν. Δεν ξέρω, θέλει κάποιον λόγο. Αν όχι, Τότε ο δόκτωρ Πρίνιε έχει τον λόγο. Φοβάμαι. Οι ερωτήσεις σας δεν είναι ακριβώς ε, ερωτήσεις. Είναι σαν ένας ε, πύραυλος με πολλούς ορόφους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος ορόφος και μετά μένει ο δορυφόρος. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Δηλαδή το επόμενο κύμα. Ειλικρινά, εγώ είμαι ιστορικός και κοιτάω το παρελθόν, όχι το μέλλον. Το μέλλον το ξέρει ο Θεός και δεν ε, είναι δική μου αρμοδιότητα. Το θέμα τώρα της βοήθειας είναι λάθος, λανθασμένο ερώτημα. Ε, θα συμφωνήσω με κάποιους που λένε ότι δεν λειτουργεί η βοήθεια. Μπορείτε να στείλετε ένα, δύο, τρία δισεκατομμύρια. Περισσότερα λεφτά για τους πολιτικούς θα είναι, θα έχουν περισσότερα λεφτά να κλέψουν. Ελάχιστα από αυτά τα λεφτά φτάνουν στους υποθέμενους δικαιούχους. Δεν είναι λύση λοιπόν. Είναι ελκυστικό γιατί ε, πατάμε ένα κουμπάκι και κάτι κάνουμε. Οπότε αισθανόμαστε ότι ε, εδώ είναι το, το πληκτρολόγιο ε, σε αντίθεση με κάτι άλλο το οποίο είναι μακριά από μένα. Αλλά το, το πληκτρολόγιο δεν είναι συνδεδεμένο με τίποτα, οπότε δεν λειτουργεί. Και νομίζω ότι έτσι, έντονες θέσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Α, ε, εντάξει, συμφωνούμε ότι ο κύριος Καμπυλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ή προσπαθούμε να τον εξαναγκάσουμε ε, κόβοντας του τη βοήθεια ξέρω για να, να αλλάξει η κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι ε, τίποτα από αυτά θα έχει αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον είναι το πώς ε, διαπραγματεύτηκαν ε, την συμφωνία της 18ης Οκτωβρίου στην Κινσάσα. Γιατί σε αυτή την κατάσταση η λύση που δεν είναι μια γενική λύση και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκων σκλαβιά και ξαφνικά είναι έτσι ωραία και ανθυρά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά η λύση είναι κάτι το οποίο προλαμβάνει μια χειρότερη καταστροφή για λίγο χρόνο έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν άλλα μέτρα. Βασικά, ο κ. Καμπυλά θα κερδίσει, θα επιβάλλει την, απόσταση, την απόφαση του, με συγχωρείτε, θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Αυτό το έχει ήδη κερδίσει. Το ερώτημα τώρα είναι να μπει κάποιος χάλινος, κάποιοι έλεγχοι στο τι μπορεί να περιμένει από την νίκη του. Γιατί η νίκη αυτή μπορεί να είναι αναποτελεσματική και να καταλήξει σε πολύ έτσι, δύσκολες καταστάσεις ή μπορεί να βγει έτσι λίγο να λειτουργεί κάπως το σύστημα. Τώρα το να χτυπάμε το χέρι μας στο τραπέζι δεν κάνει τίποτα γιατί πρέπει να στείλουμε στρατό. Αλλιώ δεν γίνεται. Το να ενθαρρύνουμε τον πληθυσμό να τον ανατρέψει είναι ανεύθυνο. Γιατί θα προσπαθήσουν. Θα προσπαθήσουν. Και μετά θα του σκοτώσουν. Και θα το κοιτάμε και θα λέμε όπω τι δραματικό, θα χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα, οι καημένοι. 200 ή 300 νεκροί το μάξιμου στις πόλεις. Ίσως και λίγο πέρα πάνω. αυτά θα είναι τα θύματα μιας τέτοιας ενέργειας να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον πληθυσμό σαν μαξιλαράκι, σαν μαξιλάρι που πετάμε δεξιά αριστερά, αυτό δεν είναι λύση. Ούτε και η βοήθεια βοηθάει. Θα ξαναγυρίσουμε σε κάτι το οποίο είναι παλιωμοδίτικο και λέγεται πολιτική. Ο Ιωσήφάκης. Έτσι το λένε ο πραγματικός ηγέτης, αυτός που έχει την εξουσία, είναι ο πατέρας Καμπυλά, όχι ο τωρινός ηγέτης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου υποστήριξη. Η υποστήριξη ερχόταν από το νότιο μέρος του Κόγκο, από την Κατάγκα και από το βόρειο και νότιο Κίβου. Τα έχει χάσει όλα αυτά. Όλη αυτή την υποστήριξη την έχει χάσει. Με τον Μπατμπόγκα τώρα έχει τον Μολουμπό ως γιατί αυτό είναι το τελευταίο ε, ψήγμα, το τελευταίο θράψμα και υποστήριξης που μπορεί να έχει και ο Μολούμπα έρχεται από το Κασάι. Η λούμπα της Κατάγκα λοιπόν τώρα έχουν στραφεί εναντίον του. Ο Κατούμι όμως δεν έχει καμιά δυνατότητα να πετύχει κάτι. Μπορεί να γίνει πρόεδρος του Κονγκό το 2025, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πολύ νωρίς για αυτόν τώρα. Θα ήταν μεγάλο το τίμημα σε ανθρώπινο αίμα. Πολιτική λύση λοιπόν σημαίνει να, να βρούμε μια ήμι πιθανότητα όπου γίνεται κάποιο άνοιγμα προς την κατεύθυνση της ε, απόδοσης της εξουσίας μετά από κάποιο εύλογο διάστημα. Αυτό δεν είναι απόλυτα ανέφικτο γιατί δεν είναι βλάκας ο πρώτος Καμπίλα, ξέρει ότι στερείται υποψή υποστήριξης, ξέρει ότι για να μείνει στην εξουσία πρέπει να σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο και αυτό θα θέσει και την περιουσία του που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, δεν ξέρω και εγώ, που αλλού στα νησιά της Παρθένου, θα κινδυνεύσουν τα λεφτά του. Αυτό το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Είναι μια διαδικασία όπου η διεθνής πίεση αυξάνεται. Θυμάμαι εποχές πανικού σε άλλες κυβερνήσεις, δεν αναφέρομαι τώρα σε ποιες, όταν κατανόησαν ότι μπορεί να βρεθούν στο σταυρόνιμα αυτών που τους ψάχνουν και τους ψάχνουν όχι να τους σκοτώσουν με όπλα, αλλά ψάχνουν τα οικονομικά τους. Επομένως ο Καμπιλά μπορεί να θέλει να μην έχει πολλούς πελάδες και θα ήθελε να έχει και κάποια επιρροή <clears throat> για το τι θα γίνει μετά ε, δεν θα μείνει για πάντα το πόλι μέχρι το 18 ή το 1919. Και αυτό είναι το σημείο που μπορεί να είναι αντικείμενο διπλωματικών συζητήσεων και επαφών, όχι για να δημιουργηθεί κάποιο πραγματικό θαύμα, αλλά για να γίνει κάτι το οποίο θα είναι <clears throat> ρεαλιστικό και εφικτό. Και υπάρχει ένας μεγάλος παίκτη σε αυτή την κατάσταση που είναι η Ρουάντα. Η Ρουάντα έχει ένα πρόεδρο που θα μείνει εκεί πέρα άλλα 25 χρόνια και θέσατε και εσείς το ερώτημα και εμεί το ίδιο, αν είναι καλή ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Αυτό που θα γίνει σε τέτοιες καταστάσεις είναι ότι απλώς κερδίζετε χρόνο. Εξασφαλίζετε την ίδια τα 5, 6, 10 χρόνια. Και όταν τα πράγματα εκραγούν, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση της ε, Ρουάντα. Εγώ ήμουν σε μια συνεδρίαση των Γάλλων Σοσιαλιστών τότε εκείνη την εποχή του πολέμου μεταξύ 1990 και της γενοκτονίας. Και η στάση της γαλλικής κυβέρνησης τότε ήταν, ήτανε υπέρ του Χαριαριμάνα λέγοντας ότι αυτό οδηγεί σε ειρήνη. Όλα πάνε καλά. Και στη συνέχεια είχαν 750.000 νεκρούς. Για μαγιά. Γιατί μετά ακολούθησαν 2,5 με 3 εκατομμύρια νεκροί στο Κονγκό. Α, οπό, οπότε κερδίζουμε χρόνο με τον κύριο Καγκαμέ. Μέχρι το 2030 θα έρθει η στιγμή να πληρώσουμε για τον χρόνο που έχουμε κερδίσει. Μπορεί να πει κανείς, όπως είπε ο Λουδοβίκος μετά από μένα, ο κατακλυσμός. Έτσι έγινε. Τότε. Με τη Γαλλική Επανάσταση που έλθε. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πάσα το θέμα στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να είναι ευνοϊκό για μας, γιατί τώρα ζούμε. <clears throat> Αν όμως είναι τα παιδιά μας που θα πρέπει να πληρώσουν για τα σπασμένα, γιατί όχι. Αλλά ούτε και αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση. Επομένως, το θέμα της διπλωματικής συζήτησης και ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κ. Κακαμέ βλέπει τι γίνεται με τον Καμπυλά. Αν τα πράγματα πάνε καλά από τη δική του άποψη, δηλαδή εμπόριο με το Κόγκο που είναι μια αγορά για τα μεταποιημένα προϊόντα της Ρουάντα, τότε θα ενισχυθεί στη θέση του. Και θα θεωρήσει ότι η διαδικασία χρονοτριβής είναι θετική γιατί της δίνει πράσινο φως η διεθνής κοινότητα. Δεν είναι λοιπόν <clears throat> μια μοναχαλήση που θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ζυγίσουμε τις μερικές λύσεις έναντι του χειρότερου σενάριου αν δεν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αν το δώσουμε βοήθεια ή να δίνουμε όπλα που δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αυτό δεν είναι λύση και ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην πολιτική όπου ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Ευχαριστώ. Κύριε Σπίλε, θέλετε να πείτε κάτι. Δεχομένως θα μπορούσα και εγώ να πω ένα-δύο πράγματα. όσον αφορά το ζήτημα της πολιτικής λύσης που θα μπορούσε να δοθεί. Δεν είναι μόνο η αλλαγή, η εναλλαγή στην εξουσία, είναι και η αλλαγή του ίδιου του συστήματος. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξεφύγουμε από προσωποπαγή συστήματα και να περάσουμε σε ένα άλλο είδος διακυβέρνησης. Θα έλεγα πάντως ότι οι τρεις μορφές αντίδρασης που ακούσαμε έχουν να κάνουν με το τρίγωνο που μας παρουσίασε ο κύριος πριν από λίγο η λέσχεση αυτή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων βλέπουμε ότι έχει και τα ωριά της σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει. Στα πλαίσια βέβαια της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν από τη γενικότερη περιφέρεια να βοηθήσουν για την πολιτική επίλυση. Έπειτα έχουμε τους ανθρώπους στο δρόμο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη ισχύ και δύναμη, αυτό βέβαια ελοχεύει κάποιου κινδύνου σίγουρα, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέρο τη απάντηση που θα δοθεί. Και η τρίτη πτυχή βέβαια είναι η διεθνή κοινότητα, εμεί. Και νομίζω ότι περιγράψαμε παρκώ τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε. Διάλογο, άσκηση πίεση, περιοριστικά μέτρα κ.ο.κ. Όσον αφορά το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τα όσα υπόθηκαν. Α μην ξεχνάμε ότι τα ποσά που έχουν ήδη εκταμιευτεί στην περιοχή αυτή ε, του κόσμου είναι τεράστια. Μιλάμε για περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ Χωρί να μετράμε καν τα χρήματα που έχουν πάει προ τη Ρουάντα. Τεράστια λοιπόν ποσά έχουν ήδη δοθεί από τη διεθνή κοινότητα. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να δούμε τώρα την ποιοτική αξιολόγηση των χρημάτων αυτών. πώ ακριβώ χρησιμοποιούνται από τα διάφορα καθεστώτα. Δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρο για την αποτελεσματικότητα ενό σχέδιου Μάρσαλ για την περιοχή όπω ακούστηκε από κάποιον. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα πολιτικά αναπτυξιακής βοήθειας, διεθνούς διπλωματίας και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, με το συνδυασμό δηλαδή όλων αυτών των εργαλείων, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια λύση, κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σπίρλετ. Κύριε Μακάιβεν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, νομίζω ότι ακούσαμε κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε απαντήσει. Όντω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δύσκολο να τανίζει κανεί το μέλλον. Αλλά μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον βασιζόμενοι στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο ήθελα και τη δική σα την συμβολή. Ξέρετε ότι το έτος 2017 θα είναι ένα πολύ σημαντικό έτος για την περιοχή αυτή της Αφρικής. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλος συνάδελφος τώρα το λόγο. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ υπάρχει κάποιος εδώ που θέλει να πάρει το λόγο. Δεν νομίζω. Είστε εδώ, είστε εδώ, λάθος, λάθος. Θέλετε παρόλα αυτά να πείτε κάτι, παρακαλώ. Έχετε, έχετε το λόγο, ενδεχομένω για τη χρηματοδότηση πείτε μας κάτι. Φραντσέσκα Ντιμάουρο από την Μονάδα Κεντρική Αφρική τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ να επιβεβαιώσω αυτό που είπε μόλι τώρα ο κύριο ε, Σπίρλετ. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουμε δώσει και για τον Μπουρούντι και για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Προφανώ αντιμετωπίσαμε δυσκολίε στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο στοχεύαμε ήταν να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντε ανάπτυξη για τι χώρε αυτέ διαχείριση των ε, φυσικών πόρων, διακυβέρνηση των φυσικών πόρων. Όλο αυτό, αυτοί οι παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη μελλοντική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Παράλληλη περιβαλλοντική προστασία, ο τομέα τη ενέργεια, ο τομέα τη υγεία. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί εκείνοι παράγοντε, οι βασικέ παράμετροι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη. Τα αναλύσαμε όλα αυτά, αλλά από μόνα του δεν αρκούν. Χρειάζεται προφανώ και πολιτική βούληση των ίδιων των κρατών αυτών για να κάνουν κάτι θετικό με τα χρήματα αυτά. Τα χρήματα πάντω υπάρχουν. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν επίσης και τα περιφερειακά ταμεία τα οποία δίδονται προς τις χώρες αυτές. Επομένω δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων σε καμία περίπτωση. Αυτό ήθελα να πω απλώς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σε ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Φοβάμαι ότι θα πρέπει όμως να κλείσουμε αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης. Θέλει κάποιο το λόγο. Συγγνώμη, δεν μπορούμε στη φάση αυτή να ακούσουμε άλλες παρεμβάσεις. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα Πρωτού περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση από την ομάδα Λευκά Κράνη. Μία ανακοίνωση πρέπει να κάνουμε, σας το συγγνώμη. So we close Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνει λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να καλωσορίσω μέλη της, του Κοινοβουλίου του Μιανμάρ, που είναι σήμερα λοιπόν εδώ παρόντα στην Επιτροπή μας. Ο κύριο Τούτουν Χέιν είναι επικεφαλής αντιπροσωπεία αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας επισκεφτήκατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.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 Υπότιτλοι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

Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτήν την δεύτερη, το δεύτερο μισό του απογεύματος. Μου ζητήθηκε να προεδρεύσω ε, εξ ονόματος του κυρίου Μπρόκ, γιατί οι άλλοι αντιπρόεδροι δεν είναι παρόντες. Θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με την ε, ομάδα πολιτικής ε, ασφάλειας στην Συρία, με τον κύριο Ραγκάλ Σελέχ, η λεγόμενη Λευκόκρανη. Η ομάδα αυτή έχει ήδη προταθεί να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, έχει υποστηριχθεί από πολλούς διεθνείς φορείς έχει βέβαια επικριθεί από φιλοκυβερνητικές οργανώσεις διότι θεωρούν ότι πρόσκειται υπερβολικά στις, στις δυτικές κυβερνήσεις. Ο κύριος Ράιτ Αλέχ, ο οποίος είναι επικεφαλής αυτού του φορέα, επρόκειτο να έρθει, αλλά τελικά δεν είναι δυνατόν να έρθει. Θα τον εκπροσωπήσουν τρεις από τους συναδέλφους, Αχμέτα Λιουσίφ, ο Αμπτούλ Ραχμάν, Αλμαουάς ο οποίος ο κύριος σύνδεσμος της οργάνωσης και ο Τζιχάντα Αλμαχαμίτ, ο οποίος είναι επίσης μέλος της οργάνωσης αυτής. Είναι γνωστή αυτή η ομάδα, ο φορέας ως Λευκόκρανη, περίπου 3.000 εθελοντές, οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι προστρέχουν για να σώσουν ζωές σε εμπόλεμες περιοχές της Συρίας. Δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας το 2013 και η χάρτα αυτής της ομάδας είναι ε, έρευνας και διάσωσης ώστε να σώσουν το μεγαλύτερο αριθμό ζώων. Είναι αμερόληπτοι, ουδέτεροι και αγωνίζονται για όλους τους Σύριους ανεξάρτητα από την ομολογία και την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Έχετε σώσει πάνω από 70.000 ανθρώπους στη Συρία και γνωρίζουμε ότι λειτουργείτε στις πιο δύσκολες συνθήκες με αυτά που γίνονται τώρα στο Χαλέπι είσαστε ήρωες της ειρήνης και η ομάδα σας, όπως ανέφερα προηγουμένως, προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ξέρουμε πόσο φρικτή είναι η κατάσταση τώρα στη Συρία και ιδιαίτερα στο Χαλέπι. Ξέρω ότι έχετε χάσει τουλάχιστον 150 εθελοντές στην περιοχή του Χαλεπίου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε στη Συρία, αλλά ιδιαίτερα και στο Χαλέπι, που φτάνει πια στο τελικό στάδιο της ε, σύγκρουσης εκεί γιατί προελάβουν οι κυβερνητικές δυνάμεις. Θα θέλαμε να ξέρουμε επίσης πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν τις προσπαθίες σας και να καλύψουν τις ανάγκες σας και να σας δώσουν <clears throat> πολιτική υποστήριξη στο έργο σας. Δίνω το λόγο για 15 λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω θα, μιλάτε, θα μιλήσετε αραβικά μέσω διερμηνίας. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο, Ιούσεφ. أشكر لكم دعوتكم لنا. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την πρόσκλησή σας. المدني السوري أو ما يسمى الخوذ البيضاء My name is Ahmed. Ahmed Al Εκπροσωπώ την ε, πολιτική προστασία της Συρίας, ε, τα λευκά κράνη. Είμαστε μια ομάδα έρευνα και διάσωσης ε, που εργάζεται για να διασώζει τραυματίες στη Συρία. Είμαστε πάνω από 3.000 εθελοντές ε, σε 120 σημεία σε 8 επαρχίες της Συρίας. Τα κέντρα αυτά είναι η ραχοκοκαλιά της δουλειάς μας. Έχουμε διασώσει μέχρι στιγμής πάνω από 73.000 ε, Σύριους και έχουμε χάσει πάνω από 150 δικούς μας εθελοντές. Οι 151 εθελοντές που χάσαμε είναι ήρωες της ανθρωπότητας και έχουμε 500 τραυματίες. Οι περισσότεροι από αυτές με μόνιμα τραύματα. Περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες ε, χτυπήθηκαν ε, στα λεγόμενα διπλά χτυπήματα. Αυτό είναι δηλαδή το χτύπημα το οποίο έρχεται 10 λεπτά μετά το πρώτο αεροπορικό χτύπημα με στόχο ακριβώς να σκοτώσει αυτούς που θα πάνε να διασώσουν. Η Συριακή κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στην έκκληση της Γαλλίας για σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ με βομβαρδισμό αμάχων. τα χτύπηματα τις τελευταίες μέρες στο Εντλίμπ και στον Κούσμα και στο Χαλέπι που σφαγιάζεται ενώπιον όλου του κόσμου. πάνω από 100 άμαχοι έχουν ε, σκοτωθεί σε αγορές ε, της πόλης ε, τις τελευταίες μέρες. Αυτό πέρα από το ότι χτύπανε σχολεία και υποδομές και νοσοκομεία. Εν ολίγης, αυτό το οποίο συμβαίνει στο Χαλέπι είναι ότι στοχεύουν τα κέντρα της ε, ζωής των αμάχων. Αυτό ακριβώς σημαίνει σε όλες τις περιοχές που είναι εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης. Και φαίνεται πως ε, το μήνυμα που θέλει να μας στείλει το καθεστώς σε μας και σε όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ότι οποιαδήποτε πρόταση για λύση δεν θα εφαρμοστεί παρά μόνο όπως θέλει το καθιστός. Και τα αποτελέσματα είναι ότι χύνεται το αίμα του Συριακού λαού. Ναι, αυτά είναι τα εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σοβαρά ε, εγκλήματα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Κυρίε και κύριοι, αυτό συμβαίνει εν ολίγη στη χώρα μου. Και ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αν ισχυρή και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει παραλύσει. Και επιτρέπει τα εγκλήματα πολέμου λόγω του βέτο της Ρωσίας. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. για να ξεφύγουμε από αυτή την διεθνή παράλυση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Συρία. για να αντιδράσουμε στους ποταμούς αίματος που χύνονται στη Συρία. Και τέλος, το μήνυμά μας σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι να σκεφτείτε την δικιά σας ανθρωπιά. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συγκινητική μαρτυρία για την ε, δουλειά που προσπαθείτε να κάνετε με τα λευκά κράνη και θέλω να πω ότι το Κοινοβουλίο έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις ακρότητες από τα αεροπορικά χτυπήματα της ε, ρωσικής ε, και της συρικής κυβέρνησης ως έγκλημα πολέμου. Ε, πραγματικά έσχος, πραγματικά αυτό το οποίο λέτε, ότι το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχει επιτρέψει κάποια ειρηνική λύση. Τόση ε, πολλοί άμαχοι έχουν πεθάνει. Εγώ προσωπικά είχα ζητήσει πριν από πέντε χρόνια μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Μου είχαν πει ότι δεν είναι δυνατόν στρατιωτικά. Έχουν χαθεί, εν πάση περιπτώσει, ε, χιλιάδες ζωές λόγω της αδράνειας της διεθνού κοινότητα. Αυτό είναι το προσωπικό μου σχόλιο, όχι ω πρόεδρο. Ο κύριο Αμπτούλ Ραχμάν ε, Αλμαχουά θέλει επίση να κάνει μια δήλωση. Έχετε τον λόγο. شكرا لكم بصراحة لم نستطع أن نرتب كلماتنا لأننا تعودنا على الفوضى في ظل ما يحدث في سوريا Thank you, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Δεν έχω προετοιμάσει κάποια δήλωση, θα ήθελα απλώς να προσθέσω κάποια σχόλια. Θα ήθελα λοιπόν να πω, ή να αναφερθώ μάλλον, σε κάποια ζητήματα πρακτικής φύσης που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα προκειμένου να βοηθηθεί η κατάσταση επιτόπου. Το 2013 επρόκειτο να επιβληθεί μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να προστατευτούν οι πολίτες, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχουμε φτάσει όμως το 2016 και αυτό που ζητούμε απλώς τώρα είναι να επιτραπεί στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στις πολιορκημένες περιοχές. Ακόμα και αν ε, η βοήθεια αυτή φτάσει εξαέρως. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, είμαστε απόλυτα σοκαρισμένοι που διεθνής κοινότητα τελικά αδυνατεί να μας βοηθήσει, αδυνατή να παράσχει βοήθεια σε μια πόλη η οποία είναι πολιορκημένη και στην οποία έχουν εγκλωβιστεί πάνω από 270.000 άτομα. Και ενώ όσο μιλάμε, η Συριακή κυβέρνηση και οι εταίροι της, οι σύμμαχοί της, συνεχίζουν και μοβαρδίζουν μια πόλη και μια περιοχή που έχει ήδη πολιορκηθεί από το Ισλαμικό κράτος. Αυτό όμω δεν μα αποσταθεροποιεί σε καμία περίπτωση. Ούτω ή άλλω δεν μπορούμε να έχουμε μια διακριτική μεταχείριση των ανθρώπων. το οποίο ζητάμε είναι τα ανθρώπινα όντα στην ε, Συρία, οι άνθρωποι στη Συρία, να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλου του υπόλοιπου ανεξαρτήτω του πού ζουν. Είμαστε βέβαιοι ότι ε, οι μελλοντικές γενιές θα αρχίσουν να αναρωτιούνται τι κάνανε άρα για την εποχή εκείνη οι ηγέτες του κόσμου για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Έχουμε φτάσει όπως σας είπα στο 2016 και σας ζητούμε για μία ακόμη φορά να βοηθήσετε τον άμαχο πληθυσμό και να επιτρέψετε στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στις πολιορκημένες περιοχές. Βρισκόμαστε εδώ τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε πεπισμένοι ότι αν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση, τότε όντως θα είστε σε θέση, θα καταφέρετε να βρείτε μια λύση. Εμείς πολλές εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσαμε να σας πούμε, δεν θα το κάνουμε αυτό τώρα, Πάντως θέλουμε να δούμε από τη δική σας την πλευρά ότι υπάρχει μια ειλικρινής πολιτική βούληση για την επίλυση της κατάστασης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημιστήριο και ο κύριος Ομπράιεν ήταν στην Επιτροπή μας την προηγούμενη εβδομάδα και κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να κινητοποιήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και για να αποτρέψουμε ε, περαιτέρω ε, επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού αλλά όπως το είπατε κι εσείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή μια συνένεση διεθνώς ανάμεσα στα διάφορα μπλεκόμενα μέρη προκειμένου να σταματήσει αυτή, αυτή η βομβαρδισμή και προκειμένου να καταλήξουμε τελικά σε μια βιώσιμη ειρήνη. Πάντως μας συγκινεί ιδιαίτερα η κατάσταση ανθρωπιστική, η ανθρωπιστική καταστροφή στη Συρία και ιδιαίτερα στο Χαλέπι. Η κυρία Μακαβάνα από την Επιτροπή Ανάπτυξης θα προεδρεύσει για τις ερωτήσεις και απαντήσεις τώρα που θα έχουμε. Νομίζω ότι ήδη θέλουν να πάρουν κάποιοι το λόγο. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω, λέει η κυρία Μακέιβεν. Όντως, πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια επί τόπου αυτό μας είπε και ο Στίβον Μπράιαν από την Ότσα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι χρειάζονται πολλές φορές έξι εβδομάδες προκειμένου να καταφέρουμε με αεροπλάνα να σας δώσουμε τη βοήθεια αυτή. Και γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκαν κιόλα και στη δυνατότητα να μπορέσουν να φτάσουν ε, με τις οδικές μεταφορές κάποιες, ε, κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Ενδεχομένως να, ε, να μπορούσατε κι εσείς να μας πείτε κάποιες πιθανές λύσεις που έχετε εντοπίσει. Κύριο Στάτινα έχει το λόγο παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ισότιμοι κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά συμπάσχω και με εσά και με τους συναδέλφους σας. Με εγγύζει ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε το γεγονός ότι έχετε χάσει τόσους πολλούς συναδέλφους σας. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ότι ε, τέτοιους ε, πολέμους έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, στη δεκαετία του 90, στην Τσέτσνια βρισκόμουν τότε, Τσετσενία με συγχωρείτε, και πραγματικά είδα εκεί με τέτοια μου τα μάτια πώς ήταν το Γκρόσνη την εποχή εκείνη. Έμοιαζε με το κομπάνι στο οποίο πήγα πέρυσι. Και όταν βλέπω εικόνες και φωτογραφίες από το Χαλέπι, Ξέρω ότι οι φωτογραφίες αυτές, οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν ακριβώς την ίδια καταστροφική κατάσταση που είχα δει και εγώ στο παρελθόν. Ας πούμε τα πράγματα επιτέλους με το όνομά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ξεκάθαρα και με απόλυτα ειλικρή, απόλυτη ειλικρίνα να πούμε τι έχει κάνει επί τόπη η Ρωσία και στην Τσετσενία, όπου δολοφόνησαν 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου και νομίζω ότι με την ίδια ειλικρίνεια θα πρέπει να μιλήσουμε και για τον βαρδισμό των Ρώσων κατά του άμαχου πληθυσμού στη δική σας τη χώρα. Και εκεί θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και θα πρέπει να καταδικαστούν βέβαια από διεθνέ δικαστήριο οι αξιωματούχοι της Ρωσίας που είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για το ηρωικό σας έργο, όλα αυτά που έχετε κάνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από πραγματικά δύσκολες και απίστευτα δύσκολες συνθήκες. Χωρίς εσάς πάρα πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν χάσει τη ζωή τους, θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερος όλεθρος ακόμα στις εμπόλεμες περιοχές, για τις οποίες εμείς δεν έχουμε κάνει και τόσο τόσα πολλά. Είναι πραγματικά είναι κάτι που θέλω να πω δημόσια. Είναι ντροπή που ο δυτικός κόσμος, ιδίως ο δυτικός κόσμος, που δίνει τόση σημασία στην προστασία των ζωών των αμάχων, δεν έχει κάνει αρκετά ή μάλλον δεν έχει κάνει τίποτα για να σας βοηθήσει. Και αυτό έχει συνεχιστεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και εμείς είμαστε απλώς στην άκρη, κοιτάμε ως θεατές και κάνουμε σαν να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε τίποτα και να βοηθήσουμε. Είναι ένας πόλεμος διαντιπροσώπων που λαμβάνει η χώρα στη Συρία. Το ξέρουμε αυτό. Και η Ευρώπη ιδιαίτερα. Θα είχε πολλά εργαλεία για να μπορέσει να χαλιναγωγήσει τις δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν εκεί γιατί έχουμε οικονομικές σχέσεις με αυτές τις χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να υποφέρουν αν εμείς σταματούσαμε το εμπόριο μαζί τους <clears throat> ως ε, τίμημα για αυτά που κάνουν στη Συρία. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ έχω σταθεί δημοσιογράφος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και έχω να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο δεν αφαιρεί τίποτα από αυτά που είπατε εσείς προηγουμένως, παρόλα αυτά θα ήθελα να το θέσω αυτό το ερώτημα. Αναρωτιέμαι πώς βλέπετε την άλλη πλευρά. Αυτούς που πολεμούν για την απελευθέρωση του Χαλεπιού, της Συρίας, ό,τι θέλουν <clears throat> τελικά να πιστεύουν. Σε ποιο βαθμό είναι υπεύθυνοι για τους πρόσθετους θανάτους που λαμβάνουν χώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει για να υπάρξει περαιτέρω ε, πίεση σε αυτές τις ε, δυνάμεις αν ελέγχονται από κάποιον εν για να προσπαθήσουν να σταματήσουν αυτή την φρικτή αιματοχυσία των πόλεμο στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασά, Μπασίρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, καθυστέρησα λίγο. Αλλά αυτά τα οποία άκουσα ήταν πολύ συγκινητικά. Σας συγχαίρω για τη σκληρή δουλειά που κάνετε και ελπίζω να συνεχίσετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής αφορά τις Ισλαμικές αξίες. Αυτά συμβαίνουν στην καρδιά του μουσουλμανικού κόσμου. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι το να αφαιρεί κανείς την ζωή ενός ανθρώπου είναι το να αφαιρεί μια, τη ζωή ενός ολόκληρου έθνους. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι όσον αφορά την μουσουλμανική διεξαγωγή του πολέμου, κατά τη διάρκεια του πολέμου που τίθεται δεν πρέπει κανείς να βλάπτει ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα λουλούδι. Τι έχει συμβεί στις μουσουλμανικές αξίες όταν έχουν σκοτωθεί 400.000 άνθρωποι μέχρι στιγμής, 7 εκατομμύρια πρόσφυγες αναζητούν προστασία σε ολόκληρο τον κόσμο, πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Θα ήθελα δεν γνωρίζω. Από θρησκευτική σκοπιά. Ε, ρωτάω γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν ε, προέρχονται από δύο πλευρές ε, του μουσουλμανικού κόσμου. Σουνίτες, Ιήτες ή κάτι άλλο και όλοι θεωρούν ότι ο Θεός είναι στο πλευρό τους. Είδαμε αυτούς τους δύο φρικτούς πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο, που όλοι έλεγαν ότι ο Θεός είναι μαζί μας τι έχει συμβεί στις μουσουλμανικές αξίες. Θα ήθελα να μάθω επειδή εσείς είστε ακριβώς στην καρδιά αυτής της υπόθεσης και το βλέπουμε κάθε μέρα. Πολλοί νέοι φεύγουν για να πάνε σε αυτόν τον πόλεμο ακούγοντας ανθρώπους που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τους λένε ότι θα κάνουν τζεχάτ και άλλες αηδίες. Εσείς είστε εκεί επί τόπου. Πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτή την ε, πραγματικά ωραία πίστη που είναι κατά της βίας. Σαλαμαλέκουμ σημαίνει έρχομαι εν ειρήνη. Λοιπόν, τι έχει πάει στραβά. Εσείς είστε επιτόπου στην Συρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Um, Κυρία Σάκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ και για την ιστορία που μας είπατε και για τη δουλειά που κάνετε. Νομίζω πως η αμεροληψία είναι μια πράξη θαραλέα την εποχή αυτή στη Συρία και το τίμημα το οποίο πληρώνεται, το, το απόλυτο τίμημα, είναι κάτι το πολύ συγκινητικό και ελπίζω να, να βρείτε στήριξη για να συνεχίσετε την δουλειά σας να βγάζετε Ζωέ από τα συντρίμια. Και παρά τις δύσκολες μέρες που περνάει η αγαπημένη σας ε, πατρίδα. Είναι ακόμη πιο οδυνηρό αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν στη Συρία τα προκαλεί ο άνθρωπος. Δεν είναι φυσική καταστροφή. Και ε, πρέπει να σα πω ότι λυπούμε και ντρέπομαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει περισσότερα για να στηρίξει τους ανθρώπους που ξεκίνησαν με ειρηνικές ε, διαδηλώσεις και ζητούσαν μια πιο ελεύθερη και δίκαιη κοινωνία, τις αξίες που υποτίθεται ότι υπερασπιζόμαστε παγκοσμίω και ε, λυπούμε για το ότι δεν υπάρχουν και περισσότεροι βουλευτές εδώ σήμερα, δεν ξέρω που έχουν πάει. Νομίζω πως όλοι θα έπρεπε να ακούσουν αυτά τα οποία είπατε. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές εδώ που μάλλον θα πούνε σκληρά λόγια στο παρελθόν είχαν στηρίξει τα καθεστώτα Πούτιν και Ασάντ και ελπίζω να μην σας ε, ενοχλήσει πάρα πολύ. Είναι η ελευθερία που έχουν οι βουλευτές, αλλά είναι μια μικρή μειονότητα που εκφράζουν. Να πω ότι ε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα πράγματα πέρα από, το, από τα λόγια και την ανθρωπιστική βοήθεια και τους πρόσφυγες ε, που προφυλάσσουμε εδώ γνωρίζοντας ότι δεν είναι αρκετά και δεν έχουμε κάνει αρκετά για να προστατεύσουμε κόσμο είτε στην περιοχή είτε μέσω της ε, Τουρκίας. Μιλήσατε για το βέτο στον ΟΗΕ και αυτό είναι πολύ προβληματικό και από Αλλά έχουμε βέτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι απίστευτο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα μια κοινή θέση για την Συρία, παρά το ότι προσπαθούμε. Και έχουμε ζητήσει κυρώσεις κατά του καθεστώτος Πούτιν που βομβαρδίζει αμάχους και σχολεία και νοσοκομεία. Και αυτό το έχει μπλοκάρει ένα βέτο της Ιταλίας, εν προκειμένου. Οπότε δικαίως απογοητεύεστε και εγώ απογοητεύομαι. Είναι απίστευτο. Και το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε και νομίζω πως αρκετοί από εμάς ε, πιέζουμε για στήριξη στην ειρηνική αντιπολίτευση, για περισσότερα μέσα και βεβαίως ε, και να ρίχνουμε και τρόφιμα από αέρος ε, και ζώνες απαγόρευσης πτήσεων έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να δολοφονούν ατιμόρυτοι μία μέρα να λογοδοτήσουν. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να γίνει αυτό. Ε, νωρίτερα, ελπίζω παρά αργότερα. Λοιπόν, ε, έχετε προταθεί για το βραβείο Νόμπελ, εγώ σας πρότεινα και για το βραβείο Ζαχάρφ και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία του χρόνου. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ τέτοιες δύσκολες μέρες. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σχάκε, εσείς ε, οργανώσατε κατά βάση αυτή την ακρόαση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που καλέσατε τους ανθρώπους αυτούς. Η κυρία Λοχπίλερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσετε το έργο σας και πραγματικά σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά αυτή που κάνετε. Προετοιμαζόμενοι για τη σημερινή συνεδρίαση, διάβασα εν συντομία τα όσα λέγονται στην ε, Wikipedia για την ε, δική σας την οργάνωση. Και υπάρχει ένας μεγάλος εκεί κατάλογος, ένας μακροσκελής κατάλογος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όντως σας υποστηρίζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν αναφέρεται η ίδια Τίθεται λοιπόν το εξή ερώτημα. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των αντίξεων αυτών συνθήκων προκειμένου να σε υποστηρίξει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της δηλαδή. Για παράδειγμα, λέτε ότι πολλοί συνάδελφοί σας έχουν ε, τραυματιστεί. Μήπως θα έπρεπε και τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τους συναδέλφους σας και να τους παρέχουν εδώ πέρα στην Ευρώπη η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και στο άρθρο αυτό της Wikipedia γίνονται και κάποιες επικρίσεις. Λέγεται ότι η Ρωσία και η Συρία σας έχουν επικρίνει γιατί λένε ότι μεροληπτείτε τελικά στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας και ότι δεν είστε ουδέτεροι. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε και αυτό παρακαλώ. Λίντα Μακέιβαν, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Επιτίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους ε, επισκέπτες μας ε, θέτοντας στο περιθώριο οποιαδήποτε πολιτική επί του θέματος θα ήθελα να σας πω ότι το έργο το οποίο επιτελείται σώζοντας ανθρώπινες ζωές είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξιέπαινο. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι δικαίως έχετε προταθεί για να λάβετε το βραβείο Νόμπελ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι εξή. Επειδή ζείτε τα πράγματα από μέσα, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να εκενωθεί ο άμαχος πληθυσμός από το χαλέπι προκειμένου, ούτως ώστε να πάψουν αυτά τα αθώα θύματα να γίνονται ανθρώπινη ασπίδα για λόγους καθαρά πολιτικούς ή όχι. Και η δεύτερη ερώτηση που έχω να σας απευθύνω είναι η εξής. Έχω ακούσει την πληροφορία ότι ο Σύριος ύποπτος για τρομοκρατία ο οποίος αυτοκτόνησε στην φυλακή στη Γερμανία ήταν μέλος της οργάνωσης σας. Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα πολωνικά και θέλω να είμαι σαφής. Σας παρακαλώ να κατανοήσετε αυτά που θέλω να πω. Εγώ χαιρετίζω την παρουσία σας και σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ εκτιμώ αυτό το οποίο κάνετε για να σώσετε ανθρώπινες ζωές. Αλλά όπως είπε και μία προλαλή σας αβουλευτής, έχετε επιτεθεί κατά του καθεστώτος του Μπασάρα Λασάντ. Ο πόλεμος, η μάχη για το Αλέπο οφείλεται στο γεγονός ότι η αντιπολίτευση, η αντιμαχόμενη των Ασάτ ή είναι χρηματοδοτούμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν είναι η αιτία του προβλήματος χρηματοδότησης αντιπολίτευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η δράση της Ρωσίας ή κάποιον άλλο. Αυτοί οι οποίοι έχουν ε, καταστήλει την ε, ε, εξέγερση στη Βαρσοβία θα πρέπει έπρεπε, θα έπρεπε να βρεθούν ενώπιον ενός δικαστηρίου, γιατί δεν επέτρεψαν στον άμαχο πληθυσμό να φύγει από την Βασοβία στην, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο ισχύει και για το Χαλέπι όμως, που κάποιοι δεν αφήνουν τον πληθυσμό, τον άμαχο πληθυσμό, να εκενώσει το Χαλέπι. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τι συμβαίνει και γιατί γίνεται αυτό, γιατί θα υπάρχουν τόση πολλά, τόσα πολλά θύματα όταν οι, οι δυνάμεις κατά του Ασάντ παραδοθούν και καταθέσουν τα όπλα. Πάντα θα πρέπει να σκεφτείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει και μία διάσωση των αμάχων. Αυτό θα πρέπει να κάνουν και οι Αμερικανοί, δεν υποστηρίζουν μόνο τις δυνάμεις κατά του, του Ασάντ. Εγώ πιστεύω ότι κάποτε θα υπάρξει η ειρήνη στην Συρία, αλλά δεν πρέπει να συνεχιστεί πολύ περισσότερο αυτός ο πόλεμος. Για μένα το απαραίτητο είναι να επανέλθει την ειρήνη και εγώ πιστεύω σε αυτά που είπε ο Ντόναλτ Τραμπ ότι δεν θα υποστηρίξει περαιτέρω τέτοιες δράσεις για να ανατρέψει δικτάτορες. Ευχαριστώ. Um, thank you, Mr. Θα μιλήσω στα, στα λετορικά. Πράγματι, οποιοδήποτε άτομο, οποιοδήποτε απλός άνθρωπος θα κατανοούσε ότι εσείς θέτετε σε κίνδυνο τη ζωή σας για να σώσετε τις ζωές άλλων ανθρώπων. Εμείς τώρα είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στις ε, στη Συρία. <clears throat> Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία μας, σε άνετες πολυθρόνες στα γραφεία μας και στις αίθουσες συνεδριάσεων. Όσα και να μας λέγατε, εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον τραγικό χαρακτήρα της κατάστασης στη Συρία. Όπως ε, είπαν κάποιοι συνάδελφοι, και αυτά μπορεί να σας φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτά. Διαβάσαμε στους New York Times ότι σας υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Βασίλειες το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι κάτω χώρε και κάποιε ΜΚΟ. Ίσως θα πρέπει να μας πείτε, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος σας δίνει χρηματοδότηση. Και επίσης σε σχέση με τον άμαχο πληθυσμό και το έργο σας. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς λειτουργείτε στις περιοχές αυτές οι οποίες είναι υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού κράτους. Πώς μπορείτε να συνεχίσετε το έργο σας όταν είναι τόσο επικίνδυνες οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι ομάδες διασωστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ήθελα να πάρω τον λόγο. Ε, ήθελα να ψηφίσω για λογαριασμό ενός συναδέλφου, αλλά ακούγοντας τους άλλους βουλευτές και επειδή γνωρίζω την δουλειά σας από την τηλεόραση, θα ήθελα να πω εδώ λίγα λόγια. Ο συνάδελφος πρότεινε μία λύση για το τι σημαίνει Συρία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κατανόηση και σεβασμό πράγματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, το, η ερώτηση για τις ε, μουσουλμανικές αξίες πρέπει να δούμε και τον ρόλο των ε, ηγετών των εκκλησιών γιατί είχα επαφή και με χριστιανούς στην Συρία και ήθελαν να, να τους βοηθήσουμε επί τόπου και μετά μας είπαν όχι, όχι, βγάλτε μας από εδώ γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Οπότε δεν ξέρω κάποιο σχόλιο για τον ρόλο των ε, επικεφαλής των εκκλησιών. Άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για απογοήτευση κτλ. Και, και συμφωνώ με τα σχόλια που είναι, ότι ε, εδώ ξέρουμε τι σημαίνει αλλά δεν το νιώθουμε και η παρουσία σας μας βοηθάει λίγο. Και πραγματικά θυμάμαι τα παιδιά που βγάζατε από τα συντρίμια, μικρά παιδιά. Και η φρίκη αυτή συνεχίζεται, οπότε θέλω και εγώ να σας στηρίξω. Ε, και είμαι απογοητευμένη που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Ε, εγώ είμαι από την Ιρλανδία. Στη Βόρεια Ιρλανδία είχαμε δύσκολο παρελθόν και ήταν δύσκολη η ειρήνη. Χρειάστηκαν προσπάθειες εκτός Ιρλανδίας. Ιρλανδίας άλλοι μας βοήθησαν έτσι ώστε στο νησί να υπάρξει ειρήνη. Αλλά εγώ γεννήθηκα σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είμαι πια νέα, αλλά χαίρομαι που τα παιδιά μου δεν βλέπουν αυτά τα οποία έβλεπα εγώ μεγαλώνοντα. Οπότε υπάρχει πάντα ελπίδα. Αν και βεβαίω ε, αυτέ τι δύσκολε στιγμέ μοιάζει να μην υπάρχει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συνάδελφοι που μου επιτρέψατε να παρέμβω σε ένα σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Δύο ομιλητέ. Έχω ακόμα. Ανελίτς πρώτα απ' όλα, του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίτς από τη Γερμανία και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχετε επαφές ε, με τους συναδέλφους. Ο Πολωνός συνάδελφος ε, έκανε μια παρομοίωση με την εξέγερση του της Βαρσοβίας ε, και είπε πως η ανθρωπιστική βοήθεια παρατείνει την κρίση. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά κρατάτε όρθιο το ανάστημα της ανθρωπότητας ε, επί τόπου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, εργάζονται εκεί επί τόπου. Συγκεκριμένη ερώτηση δική μου. Ποιες οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη σας στηρίζουν γιατί όπως είπε και η κυρία Λοχιβίλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται ε, πάρα πολύ. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα μπορούσε ίσως να ενισχύσει κάποιες από αυτές τις οργανώσεις. Σας ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος Αστοβίτσιος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όσους ε, ήρθαν και μας είπαν αυτά τα πράγματα. Ε, δύσκολο να μιλάει κανείς για την αδικία και τις κλεινοδίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν είναι κάτι το απλό. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που ακόμα ε, θέλουν να διαπράξουν τέτοια εγκλήματα και βεβαίως ε, τα εγκλήματα όταν μένουν ατιμόρυτα οδηγούν σε άλλα εγκλήματα και ε, όσοι διαπράττουν εγκλήματα ενθαρρύνονται από την παθητική θέση της ε, διεθνούς κοινότητας. Ξέρουμε τουλάχιστον δύο όνοματα, Ασάντ και Πούτιν, που ε, συνδέονται πολύ στενά. Ξέρουμε κάποιες περιφερειακές δυνάμεις επίσης που στηρίζουν και δίνουν όπλα και χρήματα σε αυτούς που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα και δεν υπάρχει αλλαγή σε αυτή την ομάδα. Θα, θα πάνε μέχρι τέλους γιατί έχουν σχέδιο. Σχέδιο το οποίο θα κοστίσει πολλές ε, ζωές και καταστροφή δυστυχώς. Ε, είναι αλήθεια. Και το βλέπουμε. Να συμβαίνει. Τα εγκλήματα λοιπόν που γίνονται και επιτοπούμε, τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ε, ζωές. Υπάρχει κάποια οργάνωση η οποία τεκμηριώνει και καταγράφει αυτά τα εγκλήματα έτσι ώστε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Υπάρχει κάποια τέτοια δραστηριότητα για την καταγραφή αυτών των εγκλημάτων και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν κάτι τέτοιο, αν κάνουν. Σας ευχαριστώ. Ακούστηκαν αρκετά πράγματα, πολλές δηλώσεις και λίγες ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Ναι, έχετε τον λόγο και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Είπατε, τι... Είπατε το τι συνέβη στο Γκρόσνη. Εγώ σπούδαζα ε, μηχανολόγος, μηχανικός ε, και, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, πραγματικά ξεπερνούν ε, το οτιδήποτε και ε, αυτά τα οποία συνέβησαν στον Κρόσνη αν δεν έχουν συμβεί στο Χαλέπι θα συμβούν στο Ιντλίμπ ε, και έχει συμβεί ήδη στα περίχωρα της Δαμασκού, στο, στη Χόμς όλοι αυτοί από εκεί εκτοπισμένοι έχουν πάει στο Ιντλίμπ οπότε έχουν φύγει να γλιτώσουν από τον δικτάτορα και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τώρα ή του χρόνου ή του παραχρόνου. Για το οικονομικό μέτωπο είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, ως ε, άμαχοι δεν νομίζω να κανείς δεν ζητάει να έρθουν άλλοι να πολεμήσουν για μας ε, κανείς δεν συμφωνεί να να πολεμήσει κάποιος άλλος για, για λογαριασμό. Τώρα υπάρχουν πολλές λύσεις οικονομικές και άλλες ε, και προς τη Ρωσία και προς το καθεστώ, για να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους και γυναικόπαιδα. Στους ε, τελευταίους ε, εκτοπισμούς είδατε τις φωτογραφίες από το Χαλέπι προς τις περιοχές που έχει το καθιστός. Οι περισσότεροι ήταν γυναικόπαιδα. Και αυτούς ακριβώς σκοτώνουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, πάνω από 200.000. Ε, πάνω από 10.000 άτομα σε δύο μέρες εκτοπίστηκαν από το Χανσί και τη Δαμασκό στο Αντλίμπ. Να σας πω λοιπόν τι συμβαίνει στο Χαλέπι. Οι δύο επιλογές έχουν οι άνθρωποι. Είτε ή θα μείνουν εκεί είτε είτε θα, πεθάνουν είτε θα, θα φύγουν. Δεν υπάρχει άλλη. Είναι σαν τους ε, βομβαρδισμούς ε, του Λονδίνου πριν από 50 ε, χρόνια ή στην Ιρλανδία Αυτό ε, ρωτάμε γιατί βεβαίω κάθε γενιά θα ερωτηθεί το, το τι έκανε. Εμεί θέλουμε να προστατεύσουμε του αμάχου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλέ πλευρέ, αλλά πεθαίνουν ε, πολλοί άμαχοι. Για την ερώτηση για τι αξίε ε, του Ισλάμ. Ευχαρίστω να συζητήσουμε τα θρησκευτικά. Πιστέψτε με, δεν έχουν αλλάξει οι αξίε του Ισλάμ. Οι μουσουλμάνοι έχουν αλλάξει. Ε, το Ισλάμ λέει ότι ε, όποιος ε, σώζει μια ζωή, σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό κάνουμε εμείς και αυτό πιστεύουμε. Για την στήριξη και το ποιος μας χρηματοδοτεί. Η USAID και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Δανία μας στηρίζουν και ε, στο επιχειρησιακό επίπεδο με εξοπλισμό, με κονδύλια, με οχήματα, με σωμικιό, με τέτοιους τρόπους και επίσης ε, για την υποψηφιότητά μας ε, για του χρόνου πραγματικά είναι πολύ ε, ευχαριστώ και είναι σημαντικό να διαδοθεί το μήνυμα μας και αν και ένας από σας πιστεύει το μήνυμα μας και μας στηρίζει Νομίζω αυτό αρκεί. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα όμως είναι δράση συγκεκριμένη για να, σταματήσει, να σταματήσουν οι θάνατοι αμάχων. Τέλος, η τελευταία ερώτηση για τα εγκλήματα πολέμου. Ε, κοιτάξτε. Είδαμε, ήμασταν μάρτυρες σε αρκετά εγκλήματα πολέμου που φορούσαν ε, την χρήση αερίου, χλωρίου, επιθέσεις σε νοσοκομεία, ε, βόμβες ε, διασποράς, ε, όλα αυτά τα στείλαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και το τελευταίο ήταν το ότι στόχευσαν βορείως του Χαλεπιού ένα ανθρωπιστικό κονβόι. Τα στοιχεία τα στείλαμε όλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά περιμένουμε. Να δούμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Αυτά. Αυτά εν ολίγης και σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος θα σας πει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ο επικεφαλής αντιπροσωπείας μάλλον θέλει να πάρει τον λόγο, αυτό είπατε τώρα. Έχετε το λόγο προφανώς, έχετε το λόγο. Η Συριακή πολιτική άμυνα δική μας θα έλεγα ότι είναι το μόνο φως σε μια κατάσταση ιδιαίτερα θλιβερή και τραγική. Είμαστε καλοί άνθρωποι, προσπαθούμε να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να μπλεκόμαστε καθόλου στην πολιτική και χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε τις πολιτικές προτιμήσεις των ανθρώπων που διασώζουμε. Μέσα σε έξι χρόνια βρισκόμαστε σε κατάσταση πραγματικής παράλυσης και εμείς να λαμβάνουμε δράση ως ασυριακή Πολιτική Άμυνα προκειμένου, διακινδυνεύοντας τη ζωή μας, να διασώσουμε ανθρώπους, ανεξάρτητα της πολιτικής κατάστασης. بيكون اسرع بالاستجابه لها لهالمناطق المكان اللي بهرب منه الناس هم بروح لعنده the areas which people... Οι περιοχές από τις οποίες φεύγει ο κόσμος εξαιτίας των ακροτήτων και των κτηνοδιών του καθεστώτος και των συμμάχων είναι οι περιοχές στις οποίες εμείς πηγαίνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα προκειμένου να σώσουμε ζωές. Ρισκάρουν λοιπόν τη ζωή τους μόνο και μόνο για να καταφέρουν να σώσουν ένα μωρό ή ένα παιδί ή μια γυναίκα από τα συντρίμια. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διακινδυνεύουν την ίδια τη ζωή τους μόνο και μόνο για να ανασύρουν τους αθώους αυτούς ανθρώπους από τα συντρίμια. بأي مشروع خلال الحرب في سوريا فهو مشروع الدفاع المدني Uh, και είναι ακριβώς αυτοί οι θεραλοί σώστε οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου για πολιτικές ατζέντε, για πολιτικές προτιμήσεις και ουσιαστικά θα θέλανε ή δυνατόν έχουν τη γενικότερη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητος προς τη Συριακή αυτή πολιτική άμυνα για να σώσουν όσο να το περισσότερες ζωές. Είμαστε περήφανοι για το έργο αυτό που κάνουμε, αλλά δεν χαιρόμαστε βέβαια που κάνουμε το έργο αυτό. Ευχόμαστε κάθε μέρα την τελευταία μέρα. يوقف Και όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, η Συριακή Πολιτική Άμυνα θα πρέπει να συνεχίσει το έργο της. Ο ήχος του όπλου, ο ήχος των βαρδισμών, καλύπτει τις φωνές των, ανθρώπων, αθώων ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε πάση θυσία τις εχθροπραξίες. Ευχαριστώ πολύ. Well, Σε ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Νομίζω ότι ακούσατε από τους συναδέλφους μας, από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πόσο θαυμάζουμε το έργο σας, με το οποίο σώζετε ζωές σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Θυμόμαστε όλοι την Τζο Κόξ, την βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες και η οποία είχε συνεργαστεί με τον φορέα σας και ήθελε να σας προτείνει για το βραβείο ειρήνης, το Νόμπελ ειρήνης. Πιστεύω ότι η Τζο Κόξ θα ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ. Θα κάνουμε λοιπόν και εγώ αρμόδια της Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω την υποστήριξή σας και ξέρω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν το ίδιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι και πάλι εξ ονόματο τη Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Θέλω και πάλι σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που είπατε και να είστε σίγουροι <clears throat> ότι μπορούμε να κάνουμε πολιτικά ή ανθρώπινα για να <clears throat> επανέλθει η ειρήνη στη Συρία θα είναι και ο στόχος μας το υπόλοιπο της εντολής μας γιατί είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αυτή η αλόγιστη αιματοχυσία, ο θάνατος τόσων αμάχων και αθώων στη Συρία. Ελπίζουμε ότι κάποτε θα επανελθεί η ειρήνη λοιπόν εκεί. Ας ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία, τις ψηφοφορίες μας για τη Συμφωνία Πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Αθενός και της Μογγολίας αφετέρου. Χέλμουτ Σόλτς είναι ο εισηγητής. Θα θέλατε να πείτε κάτι. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ενεργή τους συνεργασία. Έγιναν όλα με ένα πολύ καλό τρόπο. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Η εργασία της ε, Επιτροπής καταρχήν δεν έχει να κάνει με μια συνολική έκθεση για το, τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μογγολία, αλλά είναι πολύ καλό ότι υπάρχει αυτή η έκθεση και όλες οι πολιτικές ομάδες μπόρεσαν να συμφωνήσουν για την υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης και μετασχηματισμού της Μογγολίας. Θέλω να τονίσω επίσης ότι η Μογγολία έχει καταφέρει από μόνη της να, να χαράξει το δρόμο της παρά το γεγονός ότι έχει φυσικά ισχυρούς γείτονε όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα κατά την άποψή μας, κάτι το οποίο πρέπει να εξάρουμε στην έκθεσή μας ήταν αυτό το γεγονός. Έχουμε κάνει κάποιες συστάσεις εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει κάποια κίνηση της Μογγολίας και φυσικά τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσουν την υποστήριξή τους. Πρόκειται για θέματα όπως είναι η αηφορία και η βιωσιμότητα, αλλά και η υποστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πολιτικός διάλογος, η ανοιχτή κοινωνία. Και θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε και τη λειτουργικότητα της δημόσιας διοίκησης. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να προσθέσω, η έκθεση καταδεικνύει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις σχέσεις μας με την ε, ε, ε, Μογγολία στη σχέση μας. Εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστής των ε, γειτόνων της ε, Μογγολίας. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αμοιβαίο συμφέρον και της Μογγολίας, να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη την γραμμή που έχουν ακολουθήσει. Δεν βρήκαμε και προβλήματα εσωτερικά μέσα στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ λογικές οι συμβαστικές λύσεις και θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ λέει και ο κύριος Κέλλαμ. Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία λοιπόν. Συμβαστική τοπολογία 2. Υπέρ. Ναι, συγγνώμη. Πρώτα έχουμε το σχέδιο σύσταση όπως έχει τροποποιηθεί. Θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει, πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάω στο σχέδιο έκθεσης. <clears throat> Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάω στην τροπολογία 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εμείς χωρίς μικρόφωνο λέει ο κύριος Στάρο, θα υποστηρίσουμε όλα. Θα θέλαμε να υπάρξει μια συνολική ψηφοφορία μέχρι την ε, συμβαστική 10 αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Όχι, δεν συμφωνούν όλοι για την συμβαστική 8 είναι χωριστές ψηφοφορίες που έχουν ζητηθεί. Η ομάδα μου τις υποστηρίζει όλες. Εντάξει. Θα προχωρήσουμε, δεν χρειάζεται πολλές χώρες. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ.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 Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστές τώρα τροπολογίες. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 65 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα τη 65, υπέρ, <clears throat> κατά. Αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16. <clears throat> Έλεγχος, βεβαίως. Δεύτερο τμήμα τη 65. Πέρας. απολύθηκε πράγματι. <clears throat> Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 17 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 73 σε δύο τμήματα Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίτου. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή ας ελέγξουμε καλύτερα. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. την ψηφοφορια περας πράγματι. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. η πλειοψηφία. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 86. 86. έξι. Πέρας. απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 86. Απερίφθη. Απερίφθη. 13-13. 19. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έλεγχος για την 96 ηλεκτρονικός. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Την 8. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Σόλτς. Και έχουμε κλείσει τη συνεδρίασή μας για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους.